Right, welcome, welcome everybody. Um... Καλώς ορίσατε όλοι. Είμαι βεβαία ότι σύντομα θα χορτάσουν οι δημοσιογράφοι εδώ μπροστά, αλλά εντωμεταξύ να κλείσουμε τις διαδιπώσεις που πρέπει να γίνουν στην αρχή. Καταρχήν πρόκειται για συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών ε, Υποθέσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τα μέλη αν εγκρίνουν την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω κανέναν να είναι αντίθετος, οπότε θεωρώ πως εγκρίνεται. Θα κάνω τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχουμε συνέχιση αυτή τη συνεδρία στις 31 και περνάμε στο σημείο 3 κατευθείαν που είναι η συζήτηση για τα θέματα μακροοικονομικής πολιτικής που προκύπτουν από την τρέχουσα κατάσταση στα στο κρατικό χρέος με παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Ζαν Κλοντ Τρισέ. Να σας πω ότι πρόκειται για συζήτηση, δεν είναι ακρόαση, δεν είναι τμήμα του νομισματικού διαλόγου και είναι απαραίτητο να ακούσουμε τις απόψεις των μελών. Διάφοροι άλλοι είχαν την ευκαιρία να ακουστούν στη διάρκεια των ε, διακοπών, αλλά το Κοινοβούλιο όχι. Εν γέννη είχαμε δύσκολο καλοκαίρι. Ξέρω πως ορισμένοι από εμά δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε και όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του των θερινών διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου τα μέλη γενικώ ήταν απόντα, ενώ βέβαια κάποιοι συμμετείχαν στην ευρύτερη συζήτηση. Στόχο τη σημερινή συνεδρίαση, και ήδη είχαμε μία κυκλισμένη των θυρών συνεδρίαση με τον Πρόεδρο Τρισέ, είναι να κάνουμε μια ανασκόπηση τη τελευταία κατάσταση και να απαντήσουμε. Τι τελευταίε πέντε εβδομάδε μπορέσατε να καταλάβετε ποια είναι η αίσθηση στι χώρε σα και το να συγκεντρωθούμε ώστε να μοιραστούμε τις ε, τις συμβολές μας όλων είναι τμήμα της λύσης. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όσα έγιναν τις περασμένες εβδομάδες, εκτός το ότι να σας πω ότι ο μυθικός χαρακτήρας Sherlock Holmes είπε κάτι που θεωρώ πως είναι κέριο εδώ. Όταν δηλαδή εξαλείψεις το αδύνατο σου το απίθανο όσο απίθανο να φαίνεται. Και τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές απίθανες υποθέσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη όπως ε, τα ευρωμόλογα α πούμε που έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή. Αντίθετα όμως με το Sherlock Holmes δεν χρειάζεται να βρούμε μόνο μία απίθανη λύση, αλλά μπορεί να χρειαστούμε διάφορες απίθανες λύσεις σε στάθμη τους παράγοντες να λάβουμε υπόψη, για σε διάφορους βαθμούς μάλιστα, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πάντως, αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να εξαλείψουμε το αδύνατο, δηλαδή τον κατακαιρματισμό του ευρώ. Πολλές από τις αλλαγές που έγιναν ε, μέσω, με στόχο μάλλον ε, την αυξημένη οικονομική διακυβέρνηση πέρα από το πακέτο των έξι τη δέσμη μάλλον των έξι μέτρων μπορεί να έχουν επιπτώσεις πέρα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχει διχασμός ανάμεσα στο τι θα χρειαστεί να κάνουν ορισμένε κυβερνήσεις και το δημόσιο αίσθημα. Το να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα δεν θα το πετύχουμε με υπερβολικές ε, δόσεις ε, διακυβερνητικών διαδικασιών. Αντιθέτως, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και θα ήθελα να πω ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν πιο αξιόπιστα και συνεπή και αυτό ενισχύει την άποψή μου πως υπάρχει και ακόμα μια, ε, κάτι δεύτερο που δεν γίνεται να συμβεί, ότι το να, να σώσουμε το ευρώ να μην γίνει εις βάρος της ε, Ένωσης, της ίδιας της Ένωσης. τώρα, έχετε χρόνο δύο λεπτά έκαστος. Καταρχήν, βεβαίως θα πάρει το λόγο ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μια ενημέρωση. Και πάλι λοιπόν το λόγο έχει εσύ, Ζαν Κλοντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Χαίρομαι που σήμερα θα κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ε, μου ζητήσατε εντάχει να σας παρουσιάσω μια εικόνα των εσχάτων εξελίξεων ε, σε δημοσιοοικονομικό και νομισματικό επίπεδο στη ζώνη ευρώ, καθώς και τις πρόσφατες ε, αποφάσεις ε, σχετικά με την νομισματική ένωση. Στα γερμανικά. Από την περισμένη μας συνάντηση αυξήθηκε η σημασία ε, για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, αλλά αυτή η αύξηση ήταν επιβραδυμένη όπως είχε αν, άλλωστε κανείς περιμένει. Μεσολάβησαν πολλοί παράγοντες ε, που οδήγησαν την οικονομική ανάπτυξη τελικά να είναι μόνο ε, της τάξης του 2,2%. Αναπτύσσεται λοιπόν με μικρό ρυθμό η Ευρωζώνη, γενικά ε, σε γερές βάσεις για όλη την Ευρωζώνη. Επιπλέον, έχουν εμφανιστεί εκ νέου εντάσεις στις χρηματαγορές, γι' αυτό και είναι αρκετά μεγάλη η ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Χρειάζεται δημοσιονομική προσαρμογή σε, πολλές, ε, σε ορισμένες μάλλον από τις χώρες Ευρωζώνης, αλλά και σε άλλες αναπτυγμένες οικονομίες παγκοσμίω. Ιδιαίτερα οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, είχαν να αντιμετωπίσουν και δημοσιονομικές αλλαγές και γενικότερες μεταρρυθμίσεις σε περίοδο δύσκολη για την οικονομία. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των εμπορευμάτων και ο πληθωρισμός κινδυνεύει να αυξηθεί πάνω από 2% μέσω πρόθεσμα. Ε, υπάρχει κίνδυνος και για τη σταθερότητα των τιμών και αυτό τον καιρό το μελετούν οι υπηρεσίες μας και θα δημοσιευθεί η ανάλυση αρχές Σεπτεμβρίου. Η μεγέθυνση ε, η νομισματική παραμένει ε, περιορισμένη αλλά η ε, ρευστότητα αρκετά μεγάλη σε σχέση με ε, τις τιμές των πορευμάτων. Μάλιστα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνετοί και επιφυλακτικοί και ε, να μην χρησιμοποιείται αυτή η ρευστότητα για δαπάνες. Επιπλέον θα πρέπει να σκεφτόμαστε θερότητα των τιμών. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στην επιδείνωση των χρηματαγορών το δεύτερο ήμιση του Ιουλίου και αρχές Αυγούστου και στην Ευρωζώνη και αλλού. Στη ζώνη ευρώ εντατικοποιείται ε, η ε, μη σταθερή πορεία των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Υπάρχει μεγάλη διακύμανση των βασικών μεγεθών, κυρίως στις αγορές ε, ομολογιών. Βέβαια, πρόσφατα φαίνεται να έχει αποκατασταθεί ε, σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία τους και αν συγκρίνουμε με την κατάσταση στο Μάιο το 2010, διαπιστώνουμε ότι είναι ευρύτερη βάση λειτουργίας με πολλών αγορών πλέον και ενώπιση των εξελίξεων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει την αναχρηματοδότηση που έχει επιχειρήσει με τακτικές ε, ε, διαδικασίες τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2012. Πλήρη χρηματοδότηση, δηλαδή το σύστημα ευρώ κατοχυρώνει τι εγγύησεις ούτω ώστε να καλυφθεί η ζήτηση ρευστότητας για τις τράπεζες και να συνεχιστεί η διαδικασία αναχρηματοδότησης. Ε, η πίστη του ευρωσυστήματος στις διαδικασίες χρηματοδότησης ανέρχεται τώρα σε 530 δι ευρώ για επιχειρήσεις ε, που κυμαίνονται από μία εβδομάδα μέχρι και έξι μήνες. Αυτό το αποφασίσαμε στις αρχές Αυγούστου, δηλαδή να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία αναχρηματοδότησης και η διάρκεια κυμαίνεται περίπου ε, στις ε, έξι μήνες, ούτως ώστε να έχουν την επιθυμητή ρευστότητα οι τράπεζες. Προς το παρόν, 470 ε, τράπεζες συμμετέχουν στη διαδικασία αναχρηματοδότησης και πάνω από 600 είναι επιλέξιμες. Πάνω από 6.000 είναι επιλέξιμες. Ε, σχετικά με τους ε, τίτλους που είναι επιλέξιμοι για τις ε, διαδικασίες αυτές του στήματος ευρώ. Η αξία κυμαίνεται ανάμεσα σε 13 και 14 3 ευρώ από το, την 1η Δεκεμβρίου του 2010. Ούτω ή άλλω υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στην ετήσια έκθεση τη ΕΚΤ. Δεν υπάρχει επιλεκτική εγγύηση λοιπόν ούτε πρόβλημα με τη ρευστότητα στο συνολικό τραπεζικό σύστημα τη ζώνη ευρώ. Συνεχίζουμε τι παρεμβάσει μα ω προ τι ομολογίε, όπω αποφασίστηκε αυτό τον Αύγουστο διότι μέσα από αυτέ τι παρεμβάσει, το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΚΤ αποσκοπεί στην αποκατάσταση των προοπτικών της δημοσιονομικής και νομισματικής της πολιτικής για ε, αγορές όπου παρατηρούνται δις λειτουργίες. Δεν τροποποιείται βέβαια το νομισματικό σύστημα. Ε, συνεχίζονται αυτές οι παρεμβάσεις για να κατοχυρώσουν, όπως είπαμε, τη ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα ε, και επαναπορροφείται η ρευστότητα που προσθέτουμε στο, στο σύστημα το Μάιο του 2010 πώς είχε τοποθετηθεί η ΕΚΤ. Οι δράσεις μας ε, συνάδουν με το συνολικό στόχο της χρηματοδότησης και την εξάλληψη της ε, χρηματοπιστωτικής εξάρτησης. Ε, τα, οι ομολογίες που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις επαναγοράζονται από την ΕΚΤ στη δευτερογενή αγορά και τηρούμε τις αρχές της συνθήκης, δηλαδή η σταθερότητα των τιμών που είναι βασικός στόχος μας καθώς και κατοχυρώνουμε την ανεξαρτησία τη ΕΚ. Σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, επίση στηρούνται οι στόχοι και εφαρμόζουμε την αρχή τη αμοιβαία παρακολούθηση για τη δευτερογενή αγορά. Δεν μπορούμε τι επαναγορέ να τι χρησιμοποιήσουμε για να αναχρηματοδοτούμε την έλλειψη δημοσιονομική ε, σταθερότητα. Μοναδικό στόχο του προγράμματο είναι να διορθωθούν οι δυσλειτουργίε ε, των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η δημοσιονομική πειθαρχία έχει ε, πρωταρχική σημασία και σημειώνουμε τις επιπρόσθετες ε, διασμεύσεις που ανέβαλαν διάφορες κυβερνήσεις στη ζώνη ευρώ για να κατοχυρώσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα και την χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών. Δεν έχω λοιπόν τίποτα να τροποποιήσω σε σχέση με αυτήν την δήλωση της ΕΚΤ του Μαΐου 2010. Παραμένει έγκυρη ε, και όλοι, όλα τα κράτη, μέλη της ζώνης ευρώ εφαρμόζουν την αρχή της αμοιβαίας παρακολούθησης και τις δημοσιονομικές πειθαρχίες. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, την αυστηρή δηλαδή και έγκυρη εφαρμογή αυτών των αρχών ε, σχετικά με τα, τα πρόγραμματα προσαρμογής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Εσυνδυάζονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΚΤΕ, η έγκυρη και αυστηρή εφαρμογή της Συμφωνίας Ιουλίου 2011 ανάμεσα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης ευρώ έχει την πρωταρχική σημασία από αυτή την πλευρά. Έχει ξεκινήσει ένα ιδιαίτερο σύστημα για την Ελλάδα και ταυτόχρονα όλες οι κυβερνήσεις ε, των κρατών της ζώνης ευρώ θα μεριμνήσουν ε, ούτω ώστε να τηρηθούν οι όροι αυτής της συμφωνίας για να έχουμε ε, παρατεταμένη και βιώσιμη σταθερότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές καθώς και ως προς τη δημοσιοοικονομική διαχείριση των κρατών. Αυτά προς το παρόν, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μπορείτε και να χειροκροτήσετε, άμα θέλετε. Um, we, we to... Και ερχόμαστε τώρα στις τοποθετήσεις των Ευρωβουλευτών εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πρώτα ο κύριος Ζαν Πολ Κοζές και μετά ο Βέρνερ Λάγκεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είχα την ευκαιρία να μιλήσω προηγουμένως στη συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών, δεν θα επαναλάβω τα όσα σας είπα. Θα ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω και πάλι για την προθυμία σας να έρθετε και τον τρόπο με τον οποίο φέρεστε στους βουλευτές είναι αρκετά σημαντικό και αξίζει να σημειωθεί και δίνω το λόγο στον Βέρνερ Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στις παραμονές ε, της λήξης της ηττία σας θα ήθελα να τονίσω και εγώ ότι ανέκαθεν ε, είχατε στενές επαφές με το Κοινοβούλιο και καλλιεργούσατε ένα ειλικρινή διάλογο. Γι' αυτό χαίρομαι, γι' αυτό που είπατε, ότι στη σημερινή συνεδρίαση ε, προειδοποιείτε τις κυβερνήσεις να ασχοληθούν με την τήρηση των όσων έχουν συμφωνήσει για την εξηγήση του προϋπολογισμού και για ε, το λεγόμενο φρένο στο χρέος. Χρειαζόμαστε χρόνο στην Ευρώπη για να ε, εφαρμόσουμε τα όσα αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής. Ε, όχι μόνο ήταν σύμφωνο με το άρθρο 18 της Συνθήκης, αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ήταν υποχρεωμένη να προσφύγει στις δευτερογενείς αγορές. Και ακούγονται διάφορες επικρίσεις ε, δημοσίως, αλλά νομίζω ότι αυτή η ενέργεια ήταν απολύτως δικαιολογημένη και επιβεβλημένη θα έλεγα. Και είμαι ε, βέβαιος ότι αυτό αποδεικνύει την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ότι κάνατε αυτό το βήμα και δεν ε, δικαιώσατε τους κερδοσκόπους στις αγορές. Γιατί τις τελευταίες πέντε εβδομάδες διαπιστώσαμε ότι με φήμες και χειραγώγηση των αγορών στην περίπτωση ε, της Société Générale της Γαλλικής Τράπεζας, ε, μέσα σε λεπτά εκατοντάδες ε, εκατομμύρια κέρδισαν κάποιοι με σπέκουλα καθαρή. Και εκτός από ε, την ενίσχυση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, του πακέτου του χρηματοοικονομικού που σύντομα θα πρέπει να υιοθετήσουμε, είναι σημαντικό να σταματήσει αυτή η φόρα των αγορών Εφόσον δεν υπάρχουν ελάχιστες προθεσμίες για να διατηρεί κάποιος παράγωγα, ό,τι και να είναι αυτά, ε, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αν δεν υπάρχει λοιπόν ελάχιστος χρόνος να κρατούν στα χέρια τους οι επενδυτές αυτά τα προϊόντα, θα πρέπει να σερνόμαστε πίσω από τις αγορές. Και είναι προς τιμή σας που εσείς δεν μπήκατε σε αυτό το παιχνίδι και δεν ενδώσατε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ρητά εξ ονόματος της ομάδας μου για αυτή τη σαφή γραμμή που τηρήσατε παρόλε τι επικρίσεις που ακούτε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αν δεν είχε επέμβει η Κεντρική Τράπεζα, η ΕΚΤ, θα είχαμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι, το είπατε έμεσα, για τη ρευστότητα που δώσατε στην αγορά με ε, επαναγορά των ε, κρατικών ομολόγων. Από ό,τι κατάλαβα, ε, θα τα ξαναδώσετε πίσω όλα αυτά με ένα στοχευμένο πρόγραμμα, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά έχει χαλάσει το ρολόι. Λοιπόν θα πρέπει να δείξετε πειθαρχία όταν θα σας κάνω εγώ νοήματα. Η Ελίζα Φερέιρα από τους σοσιαλιστές παρακαλώ. Το Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που είστε και πάλι μαζί μας και σας ευχαριστώ πολύ γιατί σε διάφορα επίπεδα ξεπεράσατε την αυστηρή ερμηνεία της εντολής σας. Τούτου λεχθέντος η ισχύουσα κρίση αποδεικνύει ότι η θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η Ευρωζώνη δεν μπορεί να αντισταθεί στην ε, κρίση. Οι παρεμβάσεις γίνονται καθυστερημένα, είναι τμηματικές και η Κομισιόν δεν ανέλαβε τις ε, πρωτοβουλίες που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε και το Συμβούλιο έχει μετατραπεί σε διμερείς, μέσω μάλλον διμερών συμφωνιών, σε ένα διευθυντήριο. Εδώ εμείς προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε την κοινοτική λογική με παρεμβάσεις που βασίζονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα και όχι στην εθνική. Και Πιστεύω πως βρήκαμε μια συμφωνία με το ρόλο που θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είμαστε σε μια φάση που χρειάζεται να σκεφτούμε κάπως ευρύτερα και πιο βαθιά την υπόθεση αυτή από τον, και όχι να απαντάμε θυματικά και κατακαιρματισμένα στις διάφορες κρίσεις που ανακύπτουν κάθε τρεις και λίγο. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας ποια είναι τα στοιχεία μιας βαθύτερης, ενός βαθύτερου οράματος που από κοινού θα μπορούσαμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε την Ευρώπη σε μια προοδευτική πορεία. θα μπορέσουμε για παράδειγμα να ζήσουμε χωρίς έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας που θα είναι περισσότερο ευρωπαϊκός ε, αντί περισσότερο διακυβερνητικός και αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας μπορεί να λειτουργήσει ως, όπως λειτουργεί μέχρι στιγμής ή πρέπει να προβούμε σε αλλαγές και προσαρμογές. Μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να εκδώσουμε ευρωομόλογα. Μπορούμε να ζήσουμε με μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία θα έχει αυστηρά εντολή μόνο και μόνο τον έλεγχο των τιμών. Όταν προφανώς δεν αρκεί πια ως προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας νομισματικής ζώνης. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποια είναι η βαθύτερη δική σας άποψη, ώστε να μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε μέσω της έλλειψης πολιτικής βούλησης, αλλά και μέσω αυτού του, της έλλειψης οράματος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα εκ μέρους της ALDE. Oui, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και να θέσω μια ερώτηση. Παρατήρηση. Βλέποντας το πρόγραμμα για επαναγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και επιμένοντας και καταλάβαμε το μήνυμά σας ότι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους οι κυβερνήσεις, δεν ξεχνάμε ότι η ΕΚΤ εκπροσωπεί το ευρωπαϊκό κοινό συμφέρον και νιώθουμε ευγνώμονες και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Βεβαίως δεν μπορεί η ΕΚΤ να καλύπτει όλες τις ελλείψεις και τις αδυναμίες ε, των κυβερνήσεων. Ακολουθούσαμε μία σύγκληση με το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Ε, ήσασταν ε, στο Βερολίνο όταν η Άγγελα Μέρκελ συζητούσε τέλη Ιουλίου με τον Σαρκοζή και Αναρωτιόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο καλή την πίστη μπορούμε να ερμηνεύσουμε αισιόδοξα τις δηλώσεις τους. Ε, δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα μήνυμα για το μέλλον. Αφενός αυτές οι χώρες ε, ε, παρεμπόδισαν τις εξελίξεις στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Πώς θα γίνει τώρα οι δύο χώρες αυτές να εγκαταλείψουν τις κυρώσεις για την πλευρά της Γαλλίας σχετικά με την προληπτική υποπτία και από την πλευρά της Γερμανίας σχετικά με το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Πώς θα αλλάξουν τη στάση τους. Θα μας ε, βοηθήσετε, ούτως ώστε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, και δεν χρειάζεται τώρα να επαναλάβω αυτά που είπε η Ελίζα Φερέιρα και ο κύριος Λάγκεν, θα μας βοηθήσετε ώστε να επικρατήσει αυτό το διακυβερνητικό σύστημα, όχι με ένα άλμα ε, προς ένα ομοσπονδιακό σύστημα, αλλά χαράσοντας ε, μια ξεκάθαρη πορεία. Μπορούμε τώρα, όπως και όταν ξεκίνησε το ευρώ, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα με διάφορα στάδια καλά σταθμισμένα και έναν απότερο στόχο, ώστε οι πολίτε αλλά και οι χρηματοπιστωτικέ αγορές να καταλάβουν ότι μιλάμε και δρούμε με μία ε, φωνή. Σας ευχαριστούμε. Ε, Σουίμπερν από τους ε, συντηρητικούς. Ε, Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε Τρισέ, εδώ και δύο χρόνια ε, ανήκω σε αυτήν την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και διαπιστώνω ότι σε όλες τις παρεμβάσεις σας ε, δηλώνεται υπερήφανος και δικαίως για την ανεξαρτησία της ΕΚΤ και για τον απότερο στόχο της διατήρησης με χρηματοπιστωτικής σταθερότητα κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Και σας έχω ερωτήσει πολλά ε, Θεωρείτε χρειάζεστε περισσότερες εξουσίες στην ΕΚΤ για να μπορέσετε να παρέμβετε αποτελεσματικά στις αγορές και ανέκαθεν μας λέγατε όχι. Ε, μήπως πρέπει να τροποποιηθεί όμω η εντολή σας ε, για να μπορέσετε να εξασφαλίζετε επαρκή ρευστότητα ε, στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ και στον τραπεζικό τομέα και για να ε, αγοράζετε στις δευτερογενείς αγορές της δεκαετής ομολογίας της Ιταλίας και της Ισπανίας. Δεδομένων των διακυμάνσεων στις αγορές χρειάζεται και ένα πολιτικό κίνητρο για να μπορέσει η λειτουργία τη ΕΚΤΕ να επιδράσει αποτελεσματικά στις αγορές. Ο ρόλο τη ΕΚΤΕ είναι κέριος ε, γιατί οι πολιτικοί παράγοντες ε, δεν έχουν ε, εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του κοινού με τις δικές τους επιχειρήσεις και νομίζω ότι η ΕΚΤΑ καλείται να πάρει δύσκολες πολιτικές αποφάσεις και στις ομολογιακές αγορές δεν είναι καθόλου πεπισμένη ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια ικανοποιητική λύση. Αν δεν λοιπόν δεν έχουμε κατοχυρώσει την εμπιστοσύνη των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δεν αναγνωρίζεται η τεχνογνωσία ε, για να ε, προτείνουμε τι καλύτερε πολιτικέ ε, και τι βέλτιστε πρακτικέ. Τι προβλέπετε εσεί, μπορείτε μόλι λήξει η θητεία σα, να βοηθήσετε του πολιτικού παράγοντε και τι κυβέρνησης να λάβουν τι σωστέ αποφάσει. Νομίζω ότι οι ομολογιακέ αγορέ, οι επενδυτέ και το κοινό χρειάζεται να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη του, για να πιστούν ότι θα ανακάμψει η οικονομία και να μην βασιζόμαστε μόνο σε μη αλτρουιστέ αυτές ε, πολιτικούς. Ευχαριστούμε. Για τους πρασίνους Φίλιπ Λάμπερ. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Ε, κάποιος πράσινος, εν πάση περιπτώσει. Γκίγκολτ. Α, δεν ξέρω, δεν ε, είχαμε αποφασίσει Θέλει κάποιος θα μιλήσει. Αγαπητέ κύριε Τρισέ, φέτος το καλοκαίρι δεν ήταν τόσο χαρμόσυνο όσο περιμέναμε. Μικρότερη οικονομική ανάπτυξη, μεγαλύτερο έλλειμμα εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και έγινε και έκτακτη σύνοδος κορυφή των χωρών τη ευρωζώνη και αποφάσισαν μέτρα με εμβέλεια το πολύ δύο εβδομάδων. Και μετά χρειάστηκε να επέμβει η τράπεζα εσείς με τρόπο που σίγουρα δεν θα επιθυμούσατε αρχικά για να αναλάβετε το ρίσκο έτσι ώστε να σταθεροποιηθούν και χώρες αλλά και ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ πάρα πολύ παράδοξο και αλόκοτο τον τρόπο με τον οποίο επικρίνεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που είναι η μόνη που δρά. Επικρίνουμε αυτόν που έρχεται να σώσει αντί να λάβουμε τις ευθύνες μας. Τώρα βλέπουμε τις διάφορες χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, να ε, αναζητούν βοήθεια. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι να συμφωνήσουν 17 κοινοβούλια. Και αυτό το νέο σύστημα, το EFSF, που στο το, ε, ε, μέλλον κανονικά θα έπρεπε να σταθεροποιεί συστήματα και κράτη, δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί ε, κάθε ένα ξεχωριστό κοινοβούλιο, τώρα εθνικό, καλείται να αποφασίσει. Χρειαζόμαστε πραγματική συνεργασία στην Ευρώπη, οικονομική και μια πραγματική οικονομική ένωση και θα πρέπει να το λέμε αυτό και δημόσια και θα επιθυμούσα και ε, εσείς να κάνετε τη φωνή σας να ακούγεται δυνατά προς την κατεύθυνση αυτή και ως πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας τώρα και αργότερα. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό τώρα, πότε θα γίνει και ποιος θα το υπερασπιστεί αν δεν το πράξει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρώπη δεν πρόκειται να λειτουργήσει με μια οικονομική διακυβέρνηση από συνόδους κορυφής. Δεν γίνεται αυτό και θα καταλήξει σε αναποτελεσματική κακοφωνία και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Ο Μιγγέλ Πόρτα από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ είναι, ήθελα μόνο να πω ότι ε, όταν ο κύριος Τρισέ είπε πως δεν αποσύρει τίποτα από τα όσα είπε το 2010, εγώ θέλω να συμφωνήσω μαζί του γιατί η εισήγησή του δεν περιλάμβανε καμία καινοτομία. Αλλά υπάρχει κάτι νέο στο 2011, στο τέλη Αυγούστου που βρισκόμαστε. Η κατάσταση στην οποία ζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από οικονομική άποψη είναι πολύ χειρότερη από αυτή που επικρατούσε όταν εσείς δεν αποσύρετε τίποτα από τα όσα είπατε μέχρι τώρα. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα ότι δεν θα, δεν θα υπάρξει ανάκαμψη, δεν θα υπάρξει δημιουργία θέσεων απασχόλησης, έχουμε λιγότερη συνένεση ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά από ό,τι φαίνεται το, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι είναι σωστή, ότι δεν χρειάζεται να αναθεωρήσει τίποτα και η πραγματικότητα είναι που κάνει λάθος, όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μα δεν έχει νόημα όμω κάτι τέτοιο. Δεν έχει νόημα και θα έπρεπε και να ισχύει και κάποια ταπεινοφροσύνη. Δεν έχει γίνει καμιά αναφορά στην ευρωπαϊκή πρόταση για ομολογίες. Άκουσα να γίνεται λόγος πωλής για πληθωρισμό, αλλά δεν άκουσα μια λέξη για την απασχόληση και την ανάκαμψη της οικονομίας. Και αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα και οι προτεραιότητες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Άκουσα επίση να γίνεται λόγος για σταθερότητα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. Μα εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν δεν είχε υπάρξει δημόσια στήριξη, δηλαδή χρήματα των φορολογουμένων προς το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, πόσες ε, τράπεζες ε, θα είχαν, αντέξει τα τεστ αντοχής και μάλιστα και οι εφημερίδε λένε ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο των τραπεζών της Ευρώπης θα είχαν καταρρεύσει. Εγώ λοιπόν ανησυχώ. Ανησυχώ για τους τραπεζίτες, αλλά πολύ περισσότερο ανησυχώ για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την φρικτή κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος ε, ε, του EFT η Μάρθα Αντρίασεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, Αυξήσατε δυο φορές ε, το επιτόκιο χρηματοδότησης ε, το περασμένο χρόνο και είναι τώρα 1,5%. Ταυτόχρονα η Fed στη ΣΥΠΑ έχει φτάσει στο επιτόκιο σε 0,25% και δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να το αυξήσει. Έχουμε λάβει νέες στατιστικές από τις οικονομίες της Ευρωζώνης που δείχνουν ότι η ανάπτυξη έχει σταματήσει και ορισμένοι ειδικοί των τραπεζ... της τραπεζικής βιομηχανίας ε, βασιζόμενοι στην πρόσφατη ιστορία υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να είναι 1% κάτω από το ετήσιο ποσοστό του ΑΕΠ τα επιτόκια. Στην Αμερική ίσως αυτό να ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά στην Ευρώπη η ανάπτυξη έχει πέσει κάτω από τα επιτόκια. Ερώτημά μου είναι λοιπόν, μήπως είναι κατάλληλη στιγμή να σκεφτείτε να, να θεωρήσετε προς τα κάτω το ποσοστό επιτοκίου της ΕΚΤ, δηλαδή κατά 1% ώστε να ξεκινήσουν να κινούνται πάλι οι οικονομίες μας. Δεύτερο ερώτημα. Σχετίζεται με την κατάσταση των μεγαλύτερων οικονομιών στην Ευρωζώνη, Γερμανία και Γαλλία. Μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τις χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο, αλλά πρέπει να δούμε και την αντίδραση των ισχυροτέρων οικονομιών. Η δυσαρέσκεια είναι διαδεδομένη σε όλα τα θεσμικά όργανα και η Γαλλία δεν μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο την Ευρωσυνέλευση να συμφωνήσει για σοβαρή αντιμετώπιση του ελλείμματος. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αγνοεί αυτές τις αντιδράσεις. Σας ευχαριστώ. Χρειάζεται να συνεχίσουμε με τις παρεμβάσεις και η επόμενη από τον κύριο Μπέρχαρτ Μπέλτ του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, σας ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας. Κατά την άποψή μου η σημερινή κρίση του ευρώ δεν είναι κρίση του ευρώ ακριβώς, αλλά είναι κρίση ε, χρέους των κρατών. Γι' αυτό η απάντηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι το τέλος του ευρώ. Κατ' εμέ, ε, το θέμα είναι να λυθούν τα προβλήματα που έχουν από τα χρέη τους τα κράτη. Πολλοί λησμονούν σήμερα ότι η αλληλεγγύη μεταξύ τα κράτη-μέλη είναι βασική ιδέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Το ευρώ είναι πραγματικά η βάση της ευημερίας μας και έχουμε ζωτικό συμφέρον η νομισματική ένωση βεβαίως και να παραμείνει. Και είμαι βαθύτατα πεπισμένο ότι γι' αυτό χρειάζεται περισσότερο συντονισμό στην οικονομική πολιτική των κρατών μελών. Διότι στο μέλλον το ευρώ δεν μπορεί να είναι επιτυχές νόμισμα αν συνεχίσει να ε, αφορά 17 διαφορετικές κυβερνήσεις, 17 διαφορετικές οικονομικές στρατηγικές της κάθε χώρας. Η κρίση μας αναγκάζει να καλύψουμε το έλλειμμα του παρελθόντος που πολιτικά δεν μπορούσε να επιβληθεί ε, όταν δημιουργήθηκε το, εθνικό, το ενιαίο νόμισμα, δηλαδή με ένα συντονισμό, μια εναρμόνιση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών. Γι' αυτό καλωσορίζω τα όσα συμφώνησαν οι καγκελάριος Μέρκελ και ο Γάλλος Πρόεδρος Σάρκοζη. Μεγαλύτερος συντονισμός της οικονομικής πολιτικής και ε, ένα φρένο στο χρέος των κρατών. Αυτό το έχει ζητήσει άλλωστε και συζήτηση για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα εδώ και καιρό. Δεν θα πρέπει όμω να χάνουμε πρόφθαλμου το θέμα τη δημοκρατική νομιμότητα των αποφάσεων. Η Ευρώπη επικρίνεται πολύ σήμερα ότι είναι μακριά από τον πολίτη. Βεβαίω χρειάζεται μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό, αλλά δεν θα πρέπει να έχουν την αίσθηση οι πολίτε ότι αποφασίζουν κάποιοι ερήμην του και χωρί να του ρωτάνε τίποτα και στο τέλο καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα. Η ε, Συμφωνίε μέχρι τώρα για το συντονισμό αφορούν μόνο αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Αν θέλουμε όμω πραγματικά να έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, χρειαζόμαστε και αποτελεσματικό έλεγχο, δημοκρατικό έλεγχο τη κυβέρνηση αυτή, σε ευρωπαϊκό πάντα επίπεδο. Γι' αυτό οφείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. περισσότερη Ευρώπη για μένα δεν είναι το πρόβλημα, αλλά η λύση. Θα πρέπει όμως να βεβαιωθούμε ότι η περισσότερη Ευρώπη θα παίρνει αποφάσεις γρήγορα, αποτελεσματικά, αλλά και δημοκρατικά άψογες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες ο Ρόμπερ Γκέμπελς και δουλεύει και το ρολόι αν δεν απατώ. Ρόμπερ Γκέμπελς, ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο συνάδελφος Βένε Λάγκεν με τον οποίο συμφωνώ 100% ιδιαίτερα για την επέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη δευτερογενή αγορά. Θέλω μόνο να πω ότι ο κόσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς χρηματαγορές. Και βεβαίως αυτές οι χρηματαγορές θα πρέπει να ελέγχονται καλύτερα. Και ε, Κάπως θα πρέπει να συνεννοούνται οι οικονομικοί φορείς, αλλά ξέρουμε ότι κινούνται οι ε, ε, ρηψοκίνδυνοι traders, ας πούμε, και οι υπολογιστές τους με την ταχύτητα φωτός. Στη διάσκεψη της με, ε, η ε, Μεγάλη Βρετανία εγκατέλειψε ε, με τρόπο πάρα πολύ ηχηρό τι διαπραγματεύσει, και έλεγε στους άλλους έξι δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει αυτό που σχεδιάζεται. Ε, ε, συνέχεια τώρα μας επαναλαμβάνουν οι αγγλοσάξονες ότι το ευρώ διαλύεται. Μα το θέμα της κρίσης είναι κρίση χρέους σε ορισμένα κράτη της Ένωσης, όπως αντιμετωπίζουν αντίστοιχη κρίση πάρα πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Και κατά τη γνώμη σας κύριε Τρισέ, το ευρώ θα υπάρχει ακόμα μετά από 10 χρόνια. Πώς και είστε τόσο αισιόδοξο για το μέλλον του ευρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα τι δουλεύει το ρολόι, κάπως, σε πάση ε, από τους φιλελευθέρους, ο Ρωμόν Τρεμόζα. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Τρισέ. Καλώς ορίσατε και πάλι στο Κοινοβούλιο. Θα είμαι σύντομος. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι ακριβώς το δημόσιο χρέος της Ισπανίας που αγόρασε αυτό το μήνα η ΕΚΤ και αν υπάρχουν, ποιοι είναι οι όροι που ε, επέβαλε η ΕΚΤ στην Ισπανία για αυτήν την ε, παναγορά. Διότι έχουν καταλήξει τα ε, κόμματά μας σε μια πολύ ταχεία συμφωνία για τροποποίηση του συντάγματος. Σας ευχαριστούμε, Γαϊμό, και τώρα... Επανερχόμαστε στο ΕΛΚ. Ιωσέ Μαρία Μαγκάιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Πρόεδρε. Πολλά πράγματα συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι. Είδαμε υποβάθμιση της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Ε, είδαμε εκθέσεις που λέγουν ότι η ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι πολύ πιο ασθενής από ό,τι είχαμε προβλέψει. Με τελευταία την κυρία Λαγκάρτ να δηλώνει κάτι τέτοιο είδαμε να υπάρχουν και ε, αμφιβολίες που διασπείρονται σχετικά με το χρέος της Ισπανίας και της Ιταλίας. Και είπατε κι εσείς ότι αυτό σημαίνει 40% της Ευρωζώνης, οι χώρες που εφίστανται υποψίες από τις χρηματαγορές. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο να κάνουμε κάποιες δηλώσεις. Πρώτη, ε, δηλώσεις του κυρίου Μπερνάγκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει το επιτόκιο, θα το μειώσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να δώσει ασφάλεια στι ε, χρηματαγορές. Δεύτερον, δευτερογενής αγορά. Επανειλημμένα είπε ο κύριο Τρισέ ότι επενεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γιατί δεν μπορούσε να το κάνει κανένα άλλο, γιατί δεν εφαρμόζονται ή όσο δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις 21η Ιουλίου και επειδή ε, είχαν οδηγηθεί σε εμπλοκή κάποιες ε, καταστάσει. Και τι θα κάνει, δηλαδή ε, ε, εφόσον το Ταμείο Σταθερότητας δεν τα πράττει αυτά, θα συνεχίσει να τα πράττει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είμαι βέβαιος ε, ότι δεν θέλει να αγοράζει ομόλογα κρατικό χρέος από χώρες που δεν είναι εγγυημένο αυτό το χρέος. Εντάξει με την Ισπανία και με την Ιταλία τους στέλνει και επιστολές για να δουν τι πρέπει να κάνει για να είναι εγγυημένοι αυτή η φερεγγιότητα. Μπορείτε να μας, μπορείτε να μας δώσετε ε, τις ε, βασικές γραμμές αυτής της επιστολής, τι λέτε στις χώρες. Και μια τελευταία ερώτηση. Εγώ ανήκω στην αντιπολίτευση στη χώρα μου, αλλά η κυβέρνηση ε, έβαλε μια πιο αυστηρή οροφή στο χρέος, πιο αυστηρή ακόμα από το γερμανικό σύνταγμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ε, πραγματικά βλέπουμε μετανοημένο το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ισπανία και αυτό μας χαροποιεί. E Τώρα από το ΕΛΚ, Θεοντόρ Στολέ. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă felicit și eu, domnule președinte, al Băncii Europene. Să Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ o să να σας συγχαρώ κύριε Τρισέ, γιατί όλοι, για όλα όσα κάνατε κατά τη διάρκεια αυτού του καυτού καλοκαιριού. Χάρη στις δικές σας προσπάθειες εξευρέθη η συμφωνία για την Ελλάδα που έχει πολύ σοβαρά προβλήματα χρέους. Δεν μπορεί να βρεθεί λύση προσθέτοντας κι άλλο χρέος. Μη γίνεται λοιπόν λόγος για αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας και η ερώτησή μου είναι η εξής. Εσείς πώς ε, βλέπετε τις ενέργειες ορισμένων χωρών της, ζώνης, ε, Ευρωζώνης που θέλουν αυτή τη στιγμή να θέσουν μια ολόκληρη σειρά από προϋποθέσεις στην Ελλάδα, εγγύησεις δηλαδή, για τις οποίες δεν έγινε συζήτηση, τουλάχιστον από όσο εμείς γνωρίζουμε στη συμφωνία που επετεύχθη με την ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την λύση του προβλήματος του χρέους στην Ελλάδα. Liam, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συχνά κατηγορήθηκαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι δεν είχαν προβλέψει το πρώτο σκέλος της κρίσης. Ε, είδαμε όμως και το καλοκαίρι πόσο επιβλαβές ήταν. οι περισσότεροι που μελετούν τη συγκυρία σήμερα περιμένουν να ανατραπεί και αναθεωρούν προς τα κάτω την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και σε κάθε κράτος μέλος χωριστά. Και όλοι ανησυχούν βαθύτατα διότι η μείωση των ελλημάτων εξαρτάται από τις προοπτικές ανάπτυξης. Από την άλλη, οι τραπεζικές αξίες φέτος το καλοκαίρι ε, υπέστησαν ε, μειώσεις της τάξεως μέχρι και 40%. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σενάριο ε, με ε, μια καμπύλη που έχει σχήμα W. Και στο δεύτερο μισό λοιπόν τώρα, στο δεύτερο σκέλος, κινδυνεύουν να πέσουμε σε αυτό που κανείς δεν τολμά να αποκαλέσει ύφεση, αλλά με τεράστια ταχύτητα επιδεινώνεται η κατάσταση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπό την έννοια αυτή βεβαίω μπορεί να επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως και επενεύει, όπως είπατε προηγουμένως, ε, λάβατε αντικυκλικά μέτρα ή όπως και προτείνει ο Γκαρσία Μαργάγιο θα μπορούσε να μειώσει το διευθυντικό της επιτόκιο αλλά είναι πιθανό να βρισκόμαστε σε μια παγίδα ρευστότητα. Και υπό την έννοια αυτή και υπό τις συνθήκες αυτές δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε χωρίς δημοσιονομική πολιτική για να τονώσουμε την οικονομία ή να ανακεφαλαιώσουμε τις ε, τράπεζες, εάν αυτό ε, χρειαστεί. Θα μου πείτε δεν έχουμε περιθώριο λιγμό. Εμείς όμως οι σοσιαλιστές είμαστε οι πρώτοι που θεωρούμε ότι ένα μέγα τμήμα αυτού του χρέους ε, προήλθε από μείωση φόρων που δεν ήταν εύστοχε. Και άρα είναι αθέμητο αυτό το χρέος και εμείς θα το καταπολεμήσουμε όταν έρθουμε στην εξουσία. Έχω λοιπόν την εξή απλή ερώτηση. Στη σημερινή συγκυρία πιστεύετε σοβαρά, όπως είπατε προηγουμένως και μας καλέσατε, ότι η ενίσχυση των πολιτικών ε, εξυγίανση του προπολογισμού είναι αυτό που χρειάζεται και ιδιαίτερο στόχο στόχος του 3% για το 2013 παραμένει επίκαιρος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής από το ΕΛΚ, Κάριν Βόρτμαν Κόλ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Τρίσε, που είστε παρόν σε αυτή τη δημόσια συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι αστάθεια στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές συνεχίζεται και ότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε να βρει μια πιστική απάντηση για να λύσει το πρόβλημα χρέους και Μπορούμε να δούμε πως η οικονομική ανάπτυξη καθυστερεί λόγω όλων αυτών, σταματά. Και θα πρέπει Ίσως ε, να συνεχίσετε ναι, να, να δραστηριοποιείτε το σύστημα ε, αγοράς ομολογιών, αλλά ίσως θα πρέπει να πιέσετε και τις κυβερνήσεις ώστε να προχωρήσουν σε απαραίτητε δημοσιονομικές αλλαγές ε, και μεταρρυθμίσεις. Όπως γνωρίζετε, κάναμε πολλά με το πακέτο των έξι μέτρων. Ακούτε και την κοινή γνώμη. Υπάρχουν νέες ιδέες. Η οικονομική κυβέρνηση θα μπορούσε να αντικαταστήσει το πρόγραμμα των έξι μέτρων με πολύ ισχυρούς κανόνες που θα διέπουν αυτή τη συμφωνία. Είναι σαφές, είναι μάλλον ενδιαφέρον να ακούσουμε τη δική σας άποψη γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο μέσα στις επόμενες εβδομάδες γι' αυτό θα, ήθελα να ακούσω τα δικά σας σχόλια από αυτού. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής από το... η κυρία Ποδηματά. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε κι εσείς και πολλοί συνάδελφοι στις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου που χαρακτηρίστηκαν τότε ιστορικής σημασίας για την υπέρβαση της ε, κρίσης χρέους ε, και την ε, αντιμετώπιση της κρίσης της ελληνικής. Και σήμερα, 6-7 εβδομάδες μετά από τις αποφάσεις αυτές, όλα μοιάζουν να είναι στον αέρα και νομίζω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί. Και η δική μου απάντηση είναι ότι οι αποφάσεις εκείνες της 21ης Ιουλίου αναιρούνται σχετικοποιούνται, απειλούνται υπό το βάρος εθνικών αναγνώσεων, εθνικών ιδιαιτεροτήτων, της επικράτησης και της ονοένα και μεγαλύτερης ενίσχυσης της διακυβερνητικής προσέγγισης, για την οποία τόσα είπαμε πριν, ακόμα και εθνικών ε, αξιώσεων που παρουσιάζονται και τα οποία απειλούν συνολικά τη Συμφωνία της 21ης Ιουλίου. Και αναφέρομαι στις απαιτήσει κάποιων χωρών, κύριε Πρόεδρε, για την παροχή εμπράγματων εγγύσεων μέσω διμερού συμφωνίας προκειμένου να συμμετάσχουν στο δεύτερο πακέτο στήριξης της ε, Ελλάδας. Και πέρα από τα ζητήματα τα νομικά ή τα ζητήματα της δημοκρατίας, διότι είναι λογικό να θέλουν τα κοινοβούλια κάποιων χωρών εγγυήσεις για τη συμμετοχή των μηχανισμών του στον μηχανισμό στήριξης, αλλά είναι εξίσου λογικό ότι και τα κοινοβούλια των χωρών που δέχονται βοήθεια έχουν τα όρια τους και δεν μπορούν εύκολα να δεχθούν την υποθήκευση της χώρας τους προκειμένου να λάβουν τις εγγύσεις αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω με την ιδιότητά σας του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι ένας από τους τρεις πυλώνες των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε, το μήνυμα αξιοπιστίας για αυτά τα προγράμματα που συμφωνούμε, τα προγράμματα ε, που εκπονούνται με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Κομισιόν, όταν ζητάμε προκαταβολικά επιπρόσθετες εγγυήσεις, άρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων τελείπω αμφισβήτηση. Και κλείνω, Σάρων, Σήμερα ο Τόμας Φρίντμαν, κύριε Πρόεδρε, γράφει στη New York Times ότι η Ευρωζώνη έχει μπει σε μια διαδικασία αποσύνθεσης, διάλυσης. Εσείς μας έχετε κατ' επανάληψη τονίσει ότι δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κρίση του ευρώ, κρίση της Ευρωζώνης. Θα ήσασταν εξίσου κατηγορηματικός σήμερα όπως ήσασταν πριν από τρεις-τέσσερις μήνες. Ε, thank you. Ε, Ευχαριστούμε, Φιλίπ Λάμπερτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Σάρουν. Καλώς ορίσατε, Πρόεδρε. Η ΕΚΤ υπό την αιγίδα σας φτάνει στα όρια της εντολής της για να κατοχυρώσει τη σταθερότητα της ζώνης ευρώ και την έξοδο από την κρίση του δημοσίου χρέου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί οι όροι και προβλέπονται σε αυτή την επιστολή που έχετε στείλει στα κράτη-μέλη. Αντίθετα με αυτά που ακούσαμε εδώ όμω. δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο με μια κρίση δημοσίου χρέου, Υπαρκτή είναι, δεν πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία τη, αλλά πέρα από αυτό έχουμε μια σοβαρή κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματο στην Ευρώπη που υπερβαίνει ε, κάθε τι λογικό και η έκτη είπατε κι εσείς, ε, έχει αποφασίσει να ε, προσφέρει στο σύστημα σύστημα, ε, τη ρευστότητα, το διατραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί πλέον, οι αγορές δεν λειτουργούν πλέον και θα δώσει την απάντηση η ΕΚΤΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω, ε, σε σχέση με αυτή τη βοήθεια, ε, ποιοι είναι οι όροι που έχετε προβλέψει, δηλαδή σε σχέση με τις εγγυήσεις που θα απαιτήσετε, ποιοι είναι οι όροι που επιβάλλετε ή που θεωρείτε ότι είναι θεμητό να επιβληθούν στις τράπεζες για να αποκτήσουν την επιθυμητή ρευστότητα. Μήπως οι τράπεζες εξαρτώνται υπερβολικά από αυτό το διατραπεζικό σύστημα. Δηλαδή με συστημικό τρόπο γνωρίζετε βεβαίω ότι ε, ξεκινούμε την εξέταση τη εφαρμογή τη οδηγία Βασιλεία 3 για την Ευρώπη. Μήπω πρέπει να επιβάλλουμε μια κρίση όχι αυστηρότητα ε, αλλά μια ε, λύση περικοπών στην Ευρώπη. Μήπως πρέπει να μικρύνει το σύστημα γιατί έχει ε, επεκταθεί ε, πέραν του δέοντος. Ε, μήπως αυτό είναι το πρόβλημα του συστήματος. Ξέρουμε επίση ότι ένα κομμάτι της ρευστότητας που εσείς και άλλοι προσφέρουν στο τραπεζικό σύστημα προκύπτει από καιροσκοπικά παιχνίδια και δεν δημιουργεί καμία προστιθέμενη αξία προς την οικονομία. Ευχαριστώ τώρα η Άστρετ Λούλινγκ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε Τρισέ, θα ήθελα να σας πω πρώτα απ' όλα ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο Βένα Λάγκεν σε σχέση με το ρόλο που έχετε διαδραματίσει από το 2008 και μετά, κυρίως το 2008 όταν η Επιτροπή και το Συμβούλιο έλαμπαν δια της απουσίας τους και κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες. Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Θέλω να σας ε, ρωτήσω κάτι για την τρέχουσα κατάσταση ως προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής ε, Σταθερότητας. Ε, κατηγορούν όλοι τους πολιτικούς ότι είναι αδύναμοι ενώπιον των αγορών. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και ενισχύθηκε μετά την τελευταία σύνοδο αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, αυτό το μέσο και αυτό συνιστά μεγάλη πρόοδο κατά τη γνώμη μου. Μήπως όμως πρέπει να κάνουμε και άλλο ένα βήμα. Η αποστολή του Ταμείου ήδη διευρύνθηκε το ποσό που διαθέτει δεν επαρκεί ακόμη. Θα πρέπει να καταβάλουν και άλλες προσπάθειες ε, τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι η θεσμική πρόκληση είναι εξίσου σημαντική. Θεωρώ ότι είναι επίγον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικό Σταθερότητας ε, να εισέλθει ε, στον ευρωπαϊκό κόλπο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάγεται μόνο σε διακυβερνητικούς όρους η λειτουργία του. Δεν είναι ο στόχος του διότι είναι διακυβερνητικό αυτό το σύστημα και μακροπρόθεσμα δεν μπορεί ως εκ τούτου να λειτουργήσει. Χρειαζόμαστε ένα ουσιαστικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με κοινέ εγγυήσει για τα κράτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και όχι κατά περίπτωση να το αποφασίζουμε αυτό. Ε, δεν ξέρω αν ε, ευνοεί κάτι τέτοιο η τωρινή συγκυρία. Πώς βλέπετε εσείς την εξέλιξη, την μετεξέλιξη προς ένα ευρωπαϊκό ε, σύστημα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας τους προσεχείς μήνες, ούτως ώστε να καταδείξουμε στον κόσμο ολάκερο ότι έχουμε αναλάβει μια πλήρη δέσμευση ε, υπεράσπισης του ευρώ. Αν θεωρείτε ότι δεν είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο, θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άστριτ. Ε, Κύριε κύριος από τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τρισέ, τέλη Οκτωβρίου λέγει η θητεία σας ως Διευθυντού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αφήνετε πίσω σας ένα θεσμικό που έχει αυξηθεί σε σημασία ε, και σε επιρροή. Ποια είναι η κληρονομιά σας. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας πέρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από θεματοφύλακα σταθερότητα των τιμών να είναι ε, ο δανειστής ε, τελευταίας ε, λύσης αγοράζοντας αμφιβόλου ποιότητας ομόλογα. Κάποιοι λέγουν ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας έχει, θητεία σας έχει καταντήσει η κεντρική τράπεζα Bad Bank. Τι απαντάτε σε αυτό και τι γίνεται με την Ευρωζώνη. Σήμερα στα βιβλία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε τι ποσό έχετε κρατικά ομόλογα από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα ποσό. Ευχαριστώ πολύ. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κυρία Κράτσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπατε με μεγάλη σαφήνεια, αναφερθήκατε στο πλαίσιο της αποστολής σας για την ε, ε, προστασία του ευρώ, τη διατήρηση των τιμών ε, και επίσης για την ε, θετική εικόνα του χρηματοπιστωτικού στήματος στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σα απευθύνω δύο ερωτήσει. Πρόσφατα, η κυρία Λαγκάρτ, η Γενική Διευθύντρια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τραπεζιτών, ανέφερε ότι έκανε μια σύσταση για την κεφαλαϊκή επάρκεια των ευρωπαϊκών τραπεζών με ιδιωτικά ή δημόσια κεφάλαια συμπεριλαμβανομένων αυτών και του προσωρινού μηχανισμού στήριξης. Ε, ήθελα να σας πω πώς το κρίνετε αυτό εσείς ε, ε, για την ευρωπαϊκή ε, αγορά, τη χρηματοπιστωτική την άποψη της κυρίας Λαγκάρντ και πρόσφατα α, θα έχετε ενημερωθεί για την συγχώνευση δύο μεγάλων τραπεζών στην Ελλάδα ε, με συμμετοχή ε, 2,5 ε, δισεκατομμύρων ευρώ στο σύνολο αποκρατικό φαντ του Κατάρ. Αν αυτό δίνει μια απάντηση στο πρόβλημα ρευστότητας της Ελλάδος ή θα χρειαστούν και άλλες συγχωνεύσεις τέτοιες. Ε, και δεύτερη ερώτηση, η κυρία Λαγκάρντ στο ίδιο συνέδριο υποστήριξε επίσης ότι ο κίνδυνος της ύφεση είναι μεγαλύτερος από αυτός του πληθωρισμού και έκανε μια σύσταση πάλι για τις, την ε, προσοχή στις ε, βιαστικές δημοσιονομικές ε, προσαρμογές που εγκυμονούν κινδύνους για την ανάκαμψη. Πώς το κρίνετε αυτό εσείς κύριε Πρόεδρε και πώς βλέπετε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να συνδυαστεί με την προσπάθεια για ανάπτυξη και ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Άντελεν Σάντσες τώρα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρισέ. Και σας ευχαριστώ και για την ταχεία και αποτελεσματική δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε σχέση με τα επιτόκια, όντως η βασική σας αποστολή είναι να προσέχετε τον πληθωρισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το σημαντικότερο θέμα ο πληθωρισμός. Είναι χαμηλή η ανάπτυξη ε, και έχουμε μεγάλη διαφορά στα επιτόκια με τις ανταγωνιστικές οικονομίες και αυτό που έχει πρόβλημα τώρα δεν είναι ο πληθωρισμός αλλά η ανάπτυξη. Και για το 2013 ανακοινώνονται σενάρια χαμηλών επιτοκίων. Έχω ακούσει ήδη ε, κάποιες φήμες ε, στη Γερμανία που λένε ότι η κυρία Μέρκελ θα μειώσει τους φόρους. Δηλαδή έχουμε μια χαλαρή φορολογική πολιτική. Γιατί το κάνει αυτό. Ε, δεν χαλαρώνει την νομισματική πολιτική. Θέλει να έχει περιοριστικές πολιτικές αλλού. Ε, αλλά όταν θέλουμε περιοριστική πολιτική, όχι στο νομισματικό σκέλος, αλλά στο δημοσιονομικό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι χρέος και θα πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Το δεύτερο. Είπαμε ότι δράσατε με τρόπο ταχύ και αποτελεσματικό. Είπατε ότι ελήψη άλλων μηχανισμών θελήσατε να ε, ε, ε, παρέμβει η τράπεζα και ελπίζετε τώρα να πάρει τη σκητάλη το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Μα στην νομισματική ένωση αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε επιτόκια που να μην έχουν απεριόριστο spread. Δηλαδή για να υπάρχει νομισματική ένωση θα πρέπει να υπάρχει και ένα λογισμένο όριο και ένα οικονομικό πλαίσιο. Και αν το ορίζει το πλαίσιο ε, η κεντρική τράπεζα χάνει την εξαρτησία της. Και πώς θα το κάνει αυτό ένα ταμείο, τα κριτήρια, τα ευρωπαϊκά και η νομιμότητα. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Φιλελευθέρων Όλη Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τρισέ. Εμένα τι με ρωτάνε στην Σουηδία τακτικά. Τι κάνουν οι πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη. Κρύβονται, διακοπές είναι, πού είναι. Η πολιτική ηγεσία λείπει στην Ευρώπη και αυτό παρεμποδίζει την αίσια πορεία της Ευρώπης στο σύνολό της. Με αυτή την παρατήρηση θα ήθελα να σας χαιρετήσω από πλευράς μου και από πλευράς της ομάδας μου ε, για τον ηγετικό σας ρόλο. Δύο ερωτήσεις. Έχετε πει επανειλημμένα ότι έχουμε μια κοινή μοίρα, ένα κοινό πεπρωμένο στην Ευρώπη. Και υποθέτω ότι όταν μιλάτε για ε, τον κοινό πεπρωμένο εννοείται και τη Σουηδία και μένα. Ξέρουμε όλοι ότι 10 χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εκτός ζώνης ευρώ και φοβούμε το εξής. Μήπως διευρύνεται αυτό το χάσμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι 17 χώρες λόγω της έλλειψης ε, πολιτικής ε, ηγεσίας που κατέδειξαν σχεδόν όλες πέραν μίας ίσως, διευρύνουν αυτό το χάσμα και αυτό δεν επηρεάζει μόνο τις 17 χώρες της ζώνης ευρώ, αλλά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι πιστεύετε επ' αυτού ε, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της θητείας σας γιατί ε, ξαναλέω ότι επανειλημμένα έχετε δηλώσει πως έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο. Δεύτερη ερώτηση, αυτός ο μηχανισμός που προανέφερε η κυρία Λούλινγκ. Μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως απτή απόδειξη αλληλεγγύης μέσα στην Ευρώπη. Δεν ακριβολογούμε ή δεν ε, είναι σκόπιμο να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει ευρή ευρωπαϊκή υποστήριξη για αυτόν τον μηχανισμό. Έχει τεθεί αυτό το ερώτημα και γιατί το θέτω και εγώ, διότι θεωρώ πως ε, κάποιες χώρες εκτός Ένωσης ε, χαίρονται που είναι εκτός και όλοι επηρεάζονται από τις εξελίξεις. Όλοι, ακόμη και το ε, Ηνωμένο Βασίλειο της κυρίας Μπόλς και ε, ε, ε, ακούσατε κάπως διαφοροποιημένη τοποθέτηση του κύριο Όσμον, αλλά ακόμη και εκεί ισχύει αυτό. Καταδεικνύουμε λοιπόν ότι υπάρχει αλληλεγγύη με αυτό το μηχανισμό για τις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να δράσουμε μέσα από τον μόνιμο και προσωρινό μηχανισμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάρας από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έλεγα, κυρίες και κύριοι, δείχνει η κατάσταση ε, πόσο δύσκολη είναι. Δεν είναι καθόλου παιχνίδι αυτό που συμβαίνει. Χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα. Δεν χρειαζόμαστε μεμονωμένα εθνικά μέτρα και ε, διασφάλιση μεμονωμένων συμφερόντων, αλλά ενιαία ε, δράση με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και με πρόγραμμα. Η κρίση δεν είναι κρίση του ευρώ. Η κρίση είναι κρίση συμπεριφοράς ορισμένων πολιτικών, ανθρώπων δηλαδή που ε, προκαλούν πολιτική αστάθεια και αυτή αυξάνει την αστάθεια στις χρηματαγορές. Γι' αυτό πιστεύω ότι κανονικά θα πρέπει να κάνουμε αυτά που αποφασίσαμε, να τα εφαρμόσουμε. Το λέγανε αυτό ε, συνθήκη του Μαστρίχτ από τότε. Ε, νομισματική ένωση η οποία θα πρέπει να επιβάλλει την πολιτική ένωση. Ιδού ο στόχος μας. Δεύτερον, το ευρώ δεν διοικείται με τρόπο ε, παρέργου, δηλαδή δεν είναι παρέργο για κάποιους πολιτικούς η οικονομική διακυβέρνηση. Και είναι άλλο ένα μήνυμα ότι θέλουμε και την Ευρώπη των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Είμαστε υπέρ ε, της ευρωπαϊκής διάστασης και ενοποίησης και της κοινωνικής και, και της οικονομικής πολιτικής και της φορολογικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε οικονομική και κοινωνική ένωση, μάλιστα, και σταδιακά και βαθμιά προς τα εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Το θέμα δεν είναι το ευρώ, αλλά η αποτελεσματικότητα και η δυνατότητα δράσης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επανάκτηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης σε αυτή τη δυνατότητα λειτουργίας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σα ερωτώ, τι εννοείτε όταν λέτε ότι οι Υπουργοί Οικονομικών και οι Πρωθυπουργοί έχουν ε, την ευθύνη, την πολιτική να αναλάβουν ε, τη διακυβέρνηση του ευρώ πανευρωπαϊκά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, έξω ονόμα σοσιαλιστών και ε, δημοκρατών, ο Έντουαρτ Σικλούνα. Uh, ε, κύριε Τρισέ, στην αρχή της κρίσης ε, ακούστηκε ότι δεν είναι κρίση του ευρώ, αλλά πρόκειται για κάποιες χώρες, μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης. Αυτό υπόθηκε μετά και για τη δεύτερη χώρα. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχουν ανατραπεί τα πράγματα. Μεγάλες οικονομίες υφίστανται επιθεσει ακριβώς επειδή είναι μέλη τη Ευρωζώνης. Θα πρέπει να ε, παραδεχτούμε ότι η ίδια η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης χωλαίνει. Και το θέμα δεν είναι το ένα κράτος ή το άλλο. Θα πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα ε, δυνατό, ισχυρό, που να αντέχει σε κάποιους κραδασμούς. Χωρίς να ελαχιστοποιώ ε, τι ευθύνες των κρατών μελών, δεν πιστεύετε ότι μεταξύ ε, των εχεφρών προτάσεων είναι να υπάρχει ας πούμε ένα σύστημα αλληλεγγύης και ε, ε, μοιράσματος της ευθύνης ή του, παθητικού. Ευχαριστώ. Και τελευταίος, εξ του ΕΛΚ, τελευταία μάλλον, η κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η πρόεδρός μας άρχισε τη συνεδρίωση ε, λέγοντας ότι το να σώσουμε το ευρώ ε, μπορεί να ε, μας κοστίσει την Ευρώπη. Δηλαδή να πέσει η Ευρώπη ε, θύμα στο βωμό του ευρώ. Ανησυχώ όταν τα ακούω και δεν είμαι μόνη. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει τις ευθύνες της και κάποια άλλη, χαίρομαι γι' αυτό, ενώ ε, στα κράτη-μέλη, οι εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια πολύ συχνά κοιτούν ε, ε κοντόφλα θαλμά ε, τα δικά τους συμφέροντα. Είδαμε τι έγινε με τη δέσμη των έξι μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί, αλλά τα κράτη-μέλη διαφωνούν. Ας δούμε το μηχανισμό σταθερότητας, το έκτακτο ταμείο θα πω. Ορισμένα κράτη-μέλη αρχίζουν να ζητάνε μεμονωμένα ε, ενισχύσεις ε, και εγγυήσεις μάλλον από χώρες που θέλουν να απευθυνθούν σε αυτό το ταμείο. Ε, ζητήσαμε να υπάρχει μια κοινή βάση για το φόρο των εταιριών και για το τέλος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Έχουμε αποφασίσει κάποια μέτρα. Αν τα εφαρμόσουμε μαζί, με πίστη και με αλληλεγγύη, θα προχωρήσουμε. Έχετε και ένα μήνυμα προς τις κυβερνήσεις ε, για ε, τον τρόπο που θα πρέπει να δράσουν και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν για να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη επικάλυψη, δηλαδή κάποιες ε, ε, παρεμφερείς ερωτήσεις, ακούσαμε. Υποτίθεται ότι θα κάνουμε μία διακοπή ανάμεσα στα δύο τμήματα της συνεδρίασής μας. Ε, δεν θα γίνει διακοπή για να μπορέσουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Προσπαθήστε κύριε Τρισέ σε δέκα λεπτά να απαντήσετε σε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ήθελα να πω ότι ε, δοθείς της κατάστασης ε, δεν ξαφνιάζομαι. Με αυτές τις παρεμβάσεις άκουσα τις παρεμβάσεις, άκουσα τα πολυπληθή ερωτήματα που θέσατε. Θα προσπαθήσω ε, να είμαι σύντομος ε, στις απαντήσεις μου. Ε, από πλευράς ε, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ε, της ΕΚΤ θα ήθελα να πω το εξή ότι όλοι οι διοικητέ των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σας ευχαριστούν για τις παρατηρήσεις σας, για τα σχόλιά σας και για την αναγνώριση που μας προσφέρετε για τα όσα κάναμε τους τελευταίους μήνες. Επίσης, πολλοί βουλευτές σημείωσαν και τους ευχαριστώ ότι η πρωταρχική μας εντολή είναι να κατοχυρώσουμε την σταθερότητα των τιμών και είμαι σε θέση να σας πω ότι μετά τη θέσπιση του ευρώ το καταφέραμε αυτό, ε, τη σταθερότητα των τιμών βάσει της εντολής μας. Ε, φυσικά υπάρχει και το στοιχείο της εμπιστοσύνης, ε, δηλαδή σε θεσμικό επίπεδο υπάρχει ένα όργανο το οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε. Κάνει αυτό για το οποίο προοριζόταν και μετά από 12 χρόνια όπου ήμασταν κάτω από 2% βλέπουμε ότι σε συνολικό επίπεδο παραμένει σταθερή η κατάσταση. Αυτό που μας ζήτησαν οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες να κάνουμε νομίζω το έχουμε καταφέρει και σε κάθε δημοσκόπηση αυτό που παρατηρούμε είναι το μήνυμα που προέρχεται από τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως από τα ασθενέστερα στρώματα των συμπολιτών μας ε, που χρειάζονται περισσότερο τη σταθερότητα των τιμών ε, από ότι εμείς. Σχετικά με την ε, νομισματική πολιτική της ΕΚΤ τώρα. Ε, ό,τι κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο για να κατοχυρώσουμε τη σταθερότητα των τιμών, αυτό κάνουμε και για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις προσδοκίες όλων σχετικά με τον πληθωρισμό. Αν τώρα αυτό αντίκειται με την ιδέα ότι χρειαζόμαστε ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και πιο ενεργό δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση, εμείς θεωρούμε ότι δεν φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Ε, δεν μπορούμε να χάσουμε την εμπιστοσύνη ως προς τις προσδοκίες που υπάρχουν για τον πληθωρισμό, διότι αν συμβεί αυτό, όλα τα μακροπρόθεσμα ονομαστικά μεγέθη θα αυξηθούν, διότι ε, θα ενσωματώσουν τον επιπρόσθετο ε, πληθωρισμό που αναμένεται στο μέλλον. Δηλαδή, οι λαοί της Ευρώπης ε, θα τρομάξουν ε, διότι θα ε, διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν να εμπιστευτούν αυτό το νόμισμα που αδυνατεί να διατηρήσει την αξία του και θα εκλείψει αυτή η εμπιστοσύνη σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού πολλών χωρών και επίσης πολλών οικονομικών οργανισμών. Ε, εμείς ε, είμαστε κοντά στο 2% ή λίγο κάτω από το 2% και με αυτό τον τρόπο ε, συμβάλλουμε στην μακροπρόθεσμη ευημερία της ζώνης του ευρώ. Αυτή είναι και η βασική μας αποστολή. Ως προς την ρευστότητα τώρα, επανειλημμένα οι βουλευτές έθεσαν αυτό το ερώτημα. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο σχετικές παρατηρήσεις. Πρώτον, ε, ε, υπάρχουν κατηγορίες ότι είμαστε υπερβολικοί, ότι δίνουμε υπερβολική ρευστότητα προς τις τράπεζες και ότι δεν ελέγχουμε ε, παρκώς ε, τους εγγενείς κινδύνους αυτής της πολιτικής. Η άλλη θέση, η αντίθετη θέση είναι ότι παρά είναι ορθόδοξη η πολιτική σας, δεν προσφέρεται επαρκή ρευστότητα και δεν συνοδεύεται κατά το δέον την απαιτούμενη ανάπτυξη της οικονομίας. Εάν δούμε το σύνολο του ισοζυγίου του Ευρωπαϊκού Συστήματος, όχι μόνο της ΕΚΤ, αλλά όλων των εθνικών τραπεζών, και δούμε τι ίσχυε πριν την έναρξη της κρίσης, ας πούμε πριν από τη χρήση ε, την έναρξη των αναταράξεων, τα τέλη δηλαδή του Ιουνίου 2007 και το τι συμβαίνει σήμερα και συγκρίνω. Στη δική μας περίπτωση το ισοζύγιο, όχι μόνο της ΕΚΤ αλλά ολόκληρου του συστήματος, έχει αυξηθεί κατά 77%. Το ισοζύγιο του συστήματος ε, της ΦΕΔ έχει αυξηθεί κατά 226%. Το ισοζύγιο της ε, Κεντρικής Τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 200% και μπορώ να, σας, να συνεχίσω να σας δίνω παραδείγματα για να καταλάβετε το ότι αυτό που κάναμε είναι να κάνουμε ό,τι πιστεύουμε ότι είναι καταλληλότερο λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε με μέτρα που δεν ήταν ε, στάνταρ συμπεριλαμβανομένου του, της πλήρης, ε, χωρί, πλήρους μάλλον χορήγησης ε, ε, βοήθειας προς τις τράπεζές μας αλλά όλα αυτά έπρεπε να γίνουν με κατάλληλο προγραμματισμό και περισυλλογή για το τι είδους κινδύνους μπορούσαμε να αναλάβουμε ή όχι. Σας διαβεβαιώ λοιπόν όλους όσους πιστεύουν ότι είμαστε εξαιρετικά ε, υπερβολικά μάλλον ε, φτάρες και οι αυστηροί. νομίζω ότι δίνουμε μεγάλη προσοχή στο κίνδυνο που αναλαμβάνουμε. Και όσον αφορά τις τράπεζες ε, γενικότερα, υπόθηκαν πολλά και θα σας πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Θα έλεγα ότι μόλις, μόλις ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές αντοχής, ε, τα stress test, όλα έχουν δημοσιευθεί, είναι δυνατόν να ελέγξει κανείς συμπεριλαμβανομένων και των ε, ισοζυγίων των διαφόρων τραπεζών. Ε, των ισολογισμών με συγχωρείτε, των διαφόρων τραπεζών. Ε, έτσι μπορούν οι τράπεζες να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους με διάφορους τρόπους. Ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Βάζεις στην άκρη τα κέρδη ή βελτιώνεις, αλλάζεις τις αμοιβέ με τα πακέτα των διαφόρων συνεργατών σου. Και ένα και απαραίτητο, πας και στην αγορά και ζητάς την έκδοση και την ανακεφαλή κεφαλοποίηση νέων μετοχών και ε, πιστοτικών μέσων. Είχαμε όμως για το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα στο σύνολό του ένα τεράστιο ποσό διαθέσιμων εγγυήσεων που σαφώς υποδεικνύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλημα ρευστότητας για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του. Και πάλι έχουμε βέβαια τα μη συνηθισμένα μέτρα που σημαίνουν ότι δίνουμε ρευστότητα με σταθερό επιτόκιο, ενώ ταυτόχρονα έχουμε πολλές επιλέξιμες εγγύσεις. Σας ανέφερα τον αριθμό που είναι ανάμεσα στα 13 και στα 14, 3. Ίσως θα μπορούσα να μιλήσω και για το μέσο σταθερότητας, το οποίο γίνεται για λόγους πολιτικής ε, ε, νομισματικής. Πρέπει να γνωρίζουμε και να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η νομισματική μας πολιτική στέκει, όποια και αν είναι η άποψή μας για αυτήν, διαβιβάζεται στο σύνολο του σώματος της Ευρωζώνης σωστά. Όταν όμως δεν δυσλειτουργούν οι αγορές έχουμε πρόβλημα. Το γεγονός ότι οι αγορές δυσλειτουργούν, κατά την άποψή μας, είναι ευθύνη των κυβερνήσεων. Και από αυτού ήμουν πολύ σαφής εξασφαλίζουν τις τα δικά τους ε, χρεόγραφα, έχουν λοιπόν, εκδίδουν μάλλον τα δικά τους χρεόγραφα, τις ομολογίες τους και έχουν και την ευθύνη γι' αυτά. Φυσικά είναι προφανές ε, μεμονωμένο ότι είναι δική τους ευθύνη, αλλά εμείς θεωρούμε πως υπάρχει και συλλογική ευθύνη, διότι Ακριβώς το σύμφωνο σταθερότητας ε, υπήρχε για να ελέγχεται το τι συμβαίνει στην Ευρωζώνη και δημιουργήθηκε ακριβώς για να πούμε ότι δεν είμαστε πλήρες σε πολιτική θέση, ε, μάλλον ε, σώμα και γι' αυτό και στόχο έχουμε τον έλεγχο συλλογικά της χρήσης του δημοσίου χρήματος μέσω των δημοσιονομικών πολιτικών. Και φυσικά δεν είναι το μόνο κυβερνητικό ζήτημα που διακυβεύεται, όπως γνωρίζετε καλύτερα από όλους, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και γι' αυτό είμαστε υπεύθυνοι. Είναι, πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό στα μηνύματά μας στις κυβερνήσει. και το έχουμε πει ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν υπάρχει επιβολία από αυτό. Ακόμα και όταν δεν υπήρχαν εντάσει στην αγορά, η Ελλάδα είχε υποτίθεται τόσο αυστηρή οικονομία όσο και είπα και εν γέννη Ε, δεν είχαμε το θέμα της ε, πρακτικής της ε, αμέλειας ας πούμε, καθόλου μάλιστα και είχαμε ωστόσο το πρόβλημα όταν έπρεπε να πούμε στις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης ότι κατευθύνονται στη λάθος κατεύθυνση και ότι δεν θα πρέπει να ε, ξεπεράσετε το σύμφωνο σταθερότητας. Το 2004 και το 2005 γίνονταν αυτά. Αυτά λοιπόν για μας, εμείς θεωρήσαμε και το εξήγησε αυτό και νωρίτερα ότι υπήρχε θέμα διαβίβασης της νομισματικής πολιτικής. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να μην, να μην υπάρχει πρόβλημα ε, το μεριμνήσαμε γι' αυτό και αναμέναμε ότι και οι κυβερνήσει όπως αποφασίσαμε στις 21 Ιουλίου να προβούν στα απαραίτητα βήματα ώστε να ρυθμίσουν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσα στην Ευρωζώνη οι ίδιες οι κυβερνήσεις ε, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό και να παρεμβαίνουν στη δευτερογενή αγορά. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι ακόμα. Γενικώ το εξής. Θα πρέπει κανείς να επανέλθει στη διάσταση των ισολογισμών που σας ανέφερα. Ό,τι κάνουμε Και μάλιστα πριν από λίγο μάλιστα δημοσιεύσαμε το συνολικό ποσό της ε, παρέμβασής μας για το συγκεκριμένο πρόβλημα, για το πρόγραμμα 115 ε, δις Και αυτό που κάνουμε εδώ και λίγες εβδομάδες. Εμπαρόδο το λέγω, αλλά είναι τμήμα ε, των γενικότερων σχολείων που έκανα για τον ισολογισμό του συστήματος γενικώ. Αυτό δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν φορά μόνο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά το σύνολο των κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης. Πάρα πολλά άλλα προβλήματα επίσης εξετάστηκαν. Η διακυβέρνηση, το ε, ε, ακούσαμε γι' αυτό, είναι ένα τμήμα και ίσως το θέμα που ενδιέφερε στην αρχή τους πρώτους ομιλητές και επανήλθε πολλές φορές αργότερα στη συζήτηση. Όπως γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, γίνεται διαπραγμάτευση και θα πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα. Εμείς ζητούμε για μια πάρα πολύ σύντομη διευθέτηση. Ε, ζητούμε μια τέτοια διευθέτηση. Ήμασταν ε, στο πλευρό του Κοινοβουλίου Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, αυτό που αποφάσισαν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, ήταν να ε, ενισχύσουν τη θέση τους ως προς τη διακυβέρνηση και κατ' εμέ να έρθουν πολύ πιο κοντά προς τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα δούμε τι μέλη γενέσθε. Εγώ δεν μπορώ να υποκαταστήσω ούτε το Κοινοβούλιο ούτε τις κυβερνήσεις, αλλά εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι σημαντικό και όταν συζητούμε αυτό το θέμα της διακυβέρνησης, οφείλω να σας πω ότι για να είμαστε και ρεαλιστές, θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση αμέσως με αυτό τη λεγόμενη δέσμη των έξι μέτρων. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει. Είναι κατεπήγον και πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί. Όπως επίσης ε, σημαντικό είναι να εφαρμοστούν όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 21 Ιουλίου. Στο Άχεν εγώ μίλησα για την αυριανή ημέρα, για την επομένη και τη μεθεπομένη. Λοιπόν, υπάρχει το αύριο, υπάρχει και το μεθαύριο που θα χρειαστούν άλλες αλλαγές μεσοπρόθεσμα. Αυτά που πρόκειται να αποφασιστούν για να βελτιώσουν τη διακυβέρνηση είναι ε, δεδομένα, θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα. Γιατί, αν μου επιτρέπετε, έχουμε και την ευκαιρία, όπως κάθε προηγμένη οικονομία να κάνουμε μια ακτινογραφία ε, στην Ευρωζώνη, στα 17 κράτη. Αλλά δεν είναι μόνο Αυτό είναι μια από τις χειρότερες κρίσεις ε, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ίσως η χειρότερη και θα το τολμούσα να πω ότι ενδεχομένω αν δεν είχαμε αντιδράσει εγκαίρως να ήταν και η χειρότερη κρίση από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μιλώ για τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, τέτοιες κρίσεις συμβαίνουν κάθε 60-70 χρόνια. Δεν έχει περάσει, είναι ένα συνεχιζόμενο φαινόμενο, έχει αποκαλύψει κάποιες αδυναμίες και στις Ηνωμένες και στην Ιαπωνία και στην Ευρώπη και αυτό δεν μας και θα πρέπει να βγάλουμε όλα τα συμπεράσματα που ε, ζητούν διαρθρωτικές αλλαγές. Και απηχώ και εγώ και συμφωνώ με ε, πολλά από όσα είπαν πολλοί βουλευτές για τη ε, διάσταση αυτή τη διαρθρωτική για το αύριο, αλλά το σήμερα απαιτεί να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε αποφασίσει σήμερα και να αποκρισταλωθούν στην πράξη αυτά που διαπραγματευθήκαμε για τη διακυβέρνηση και οι αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε αρκετή γενναιοδορία για να μου δώσετε και άλλο χρόνο. Ε, έχω ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο που μου δώσετε, με μεγάλη γενναιοδορία όντως, αλλά πρέπει να σας πω το εξής. Είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θέλουμε να υπερβούμε καθόλου ευθύνη μας και το ρόλο. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίζουμε τη σταθερότητα των τιμών. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό το κάναμε. Και αυτή τη στιγμή που σα μιλώ, ακόμα και μέσω αυτής της κρίσης, θα φερέγγιοι και αξιόπιστοι ε, από όλους τους ε, φορείς και τους συμμετέχοντες της αγοράς για την επόμενη δεκαετία, ότι είναι δεδομένη ε, σταθερότητα. Και αυτό πραγματικά ε, πιστώνεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι πάρα πολύ σκληρή ε, ε, καιρή για μας, όπως και για όλες τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις. Αυτό που κάνουμε είναι μόνο μέσω από το πρίσμα της νομισματικής πολιτικής, γιατί αυτή είναι η ευθύνη μας, να παίρνουμε τις αποφάσεις όταν χρειάζεται ε, για την νομισματική πολιτική, για λόγους νομισματικής πολιτικής και να στέλνουμε μηνύματα σε κυβερνήσεις σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο ε, της Ευρωζώνης στο σύνολό της, δηλαδή τι αντίκτυπο θα έχει η λήψη αποφάσεων ή η μη λήψη αποφάσεων από πλευρά του σε όλη την Ευρωζώνη. Πρόσφατα είχαμε επαφές με τις κυβερνήσεις, στέλνουμε λοιπόν μηνύματα, όντως, δεν διαπραγματευόμαστε, μηνύματα απευθύνουμε και είπαμε ότι αν θέλουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη που έχει κλονιστεί σε μεγάλο βαθμό, κατά την άποψή μας ε, χρειάζεται να λάβετε τα εξή μέτρα ή να πάρετε τον εξή ε, προσανατολισμό. Χωρίς διαπραγμάτευση. Όταν όμως έλαβαν τις αποφάσεις ακριβώς επειδή είχαν κατανοήσει πλήρως ότι χρειάζεται να επανέλθει η εμπιστοσύνη της υπογραφής. Ε, λήφθησαν οι αποφάσεις λοιπόν μετά ε, από εξέταση των όσων αποφασίστηκαν. Δεν ήταν διαπραγμάτευση, επαναλαμβάνω. Μηνύματα στέλνουμε. Και είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε ε, απολύτως και να το κατανοούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, τα θα τα καταφέρετε τώρα να δραπετεύσετε και να αφήσετε τη θέση στον επόμενο στο διάδοχό σας ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σούσεις της κρίσης. Ε, καλή τύχη, σας ευχαριστούμε. Έχουμε ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα. Ουσιαστικά δεν έχουμε κανένα διάλειμμα. Right, Καθίστε παρακαλώ όλοι. Ώστε, μόλις πιάσω τον Υπουργό, να ξεκινήσουμε. Would stop ναι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. much um, Σας ευχαριστώ όλους. Όπως γνωρίζετε έχουμε μια κάποια καθυστέρηση, αλλά ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα όσα έχουμε προβλέψει. Ερχόμαστε στη δεύτερη συζήτηση που είναι η συζήτηση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνη στην αγορά, νομοθετικές και θεσμικές απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι μαζί μας ο, ο Υπουργός που είναι προεδρεύων του Συμβουλίου από την Πολωνία. Έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Ζαν Πολ Γιούγκερ και τον Επίτροπο για τα Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα, τον Όλη Ρεν. Και με αυτή τη σειρά θα πάρουν το λόγο. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω δηλώσεις που έκανα στην έναρξη αυτής της συνεδρίασης. Διαβίβασα τα σχόλιά μου στους ομιλητές χωρίς άλλη καθυστέρηση και αν θα μπορούσαν ε, και οι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης να φύγουν σιγά σιγά εδώ από μπροστά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στον Υπουργό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τιμή μου και προνόμιό μου να είμαι σήμερα εδώ ενώπιόν σας καθώς προεδρεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είδαμε την ταχύτητα με την οποία η κρίση μπορεί να βαθύνει και να αναπτυχθεί. Η ευρωπαϊκή κρίση δηλαδή της Ευρωζώνης. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό για μας ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο να μπορέσουμε να αναλύσουμε σωστά τους λόγους που κρύβονται πίσω από την κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και έτσι να καταφέρουμε να βρούμε και κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα αυτά. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενος στο προηγούμενο τμήμα της συζήτησης με τη συμμετοχή του Προέδρου της ΕΚΤ, κ. Τρισέ. Και εδώ θα ήθελα να πω τα εξής. Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τον Αύγουστο Κατά τη γνώμη μου και χωρίς καμία επιφύλαξη ή αμφιβολία και το λέω αυτό με πλήρη συνέστηση των λόγων μου, οι ενέργειες της ΕΚΤ κατάφεραν να σώσουν την Ευρώπη. Νομίζω πως οποιαδήποτε αμφιβολία ή δισταγμός από πλευράς της ΕΚΤ θα μπορούσε να έχει καταλήξει κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα σε μια πολύ χειρότερη κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι ενέργειες τις οποίες προέβη η ΕΚΤ ήταν ε, οι σωστές και πλήρως ευθυγραμμισμένες με την, νομική, με την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και όχι μόνο ήταν νόμιμες και ήταν και νόμιμες τότε που έγιναν οι ενέργειες αυτές, αλλά ήταν και απολύτως απαραίτητες. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός αυτό και πραγματικά να εκτιμούμε τις ενέργειες της τράπεζας και του Προέδρου της. Ως Ευρώπη έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ στον ομιλία του στο Στρασβούργο πριν ε, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε σαφώς ότι χωρίς αλληλεγγύη η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Και νομίζω πως αυτό το διαπιστώνουμε σήμερα. Μόλις 6-7 εβδομάδες αργότερα από την ομιλία αυτή του Πολωνού Πρωθυπουργού αντιμετωπίζουμε Έχουμε μάλλον να προβούμε σε μια επιλογή. Απ' τη μια είναι η αλληλεγγύη, απ' την άλλη η κατάρρευση της Ευρώπης. Φυσικά αυτή η αλληλεγγύη απαιτεί την συνειδητοποίηση των συμφερόντων μας. Οι χώρες με πλεόνασμα θα πρέπει αυτό να το, να το αναγνωρίσουν, δηλαδή ο πλούσιος βορράς εντός της Ευρωζώνης, αλλά και η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνει κατανοητή από πλευράς των νοτίων χωρών ή και κάποιων χωρών που βρίσκονται σήμερα σε προβληματική κατάσταση. Αλλά γνωρίζουμε πως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της αλληλεγγύης, ότι αν δηλαδή βοηθήσουμε κάποιον σήμερα, τότε στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον ίσως, θα το ανταποδώσει και μάλιστα με τόκο. Ε, επιπλέον αυτή η αλληλεγγύη είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των όσων παίρνουν τη βοήθεια αλλά και των όσων την παρέχουν. Να αναφέρω ένα θέμα κλειδί. Την δέσμη των έξι ε, μέτρων που αυτή τη στιγμή συζητάται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κατά τη γνώμη της Πολωνικής Προεδρίας, η κατάσταση είναι τέτοια που ευερετέρω ολοκλήρωση είναι απαραίτητη σήμερα και ε, μακροοικονομικά αυτή η ολοκλήρωση είναι απαραίτητη για τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτή η περαιτέρω λοιπόν ολοκλήρωση θα πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό κοινοτική φύσης. Και η Πολωνία, ως χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης, θεωρεί πως είναι εξαιρετικά σημαντικό η... να προχωρήσει η ολοκλήρωση επί τη βάση των κοινοτικών αρχών. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε πως η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη είναι τόσο σοβαρή που ε, αν εμείς ως ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δηλαδή Συμβούλιο, Κομισιόν, Κοινοβούλιο, αν δεν καταφέρουμε να αποδείξουμε στην υπόθεση του πακέτου των έξι μέτρων ότι είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε γρήγορα κοινή θέση και να εφαρμόσουμε τα μέτρα αυτά σύντομα και γρήγορα, τότε είτε το θέλουμε είτε όχι, τα κράτη-μέλη θα αναγκαστούν να βρουν διαφορετικές λύσεις. Ενώπιον αυτής της σοβαρής απειλής, την οποία αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ευρωζώνη, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη, η Πολωνία ως κράτος μέλος που είναι απόλυτα πεπισμένο για την ορθότητα της κοινοτική μεθόδου θα ήθελε να τονίσει ότι το θέμα του πακέτου των 6 μέτρων θα είναι ένα τεστ αντοχής για όλους μας. Για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι μια δοκιμασία για το κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κοινοτική μέθοδο για να ενεργήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό, ας μην τρέχουμε αφιβολίες. Οι λύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν δεν θα είναι κοινοτικέ μετά, γιατί αυτό θα σημαίνει πως η κοινοτική μέθοδος θα έχει αποτύχει σε τόσο δύσκολους καιρούς. Κάτι ακόμα να σας πω. Να προσθέσω λοιπόν ότι οι ειδικοί αναλυτές, ιδιαίτερα στην ε, χρηματοπιστωτική αγορά, λένε ότι οι περαιτέρω προσαρμογές και περαιτέρω περιορισμός των ε, ε, προσαρμογών και μάλλον της ανάπτυξης παγκοσμίω είναι αυτό που μας περιμένει. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να αυταπατώμεθα ένα μεγάλο τμήμα αυτής της ύφεσης, της αναμενόμενης ύφεσης, προκύπτει από αυτήν την ε, πολιτική αβεβαιότητα που περιβάλλει την Ευρωζώνη και το πακέτο των έξι πολλοί κόσμος διστάζει για να επενδύσει σε νέα σχέδια και νέες θέσεις απασχόλησης, γιατί γνωρίζει ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την σταθερότητα της Ευρώπης, απειλές που προκύπτουν από το πακέτο. Να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν λαμβάνουμε πάντοτε αποφάσεις αρκετά γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο είμαι πεπισμένος ότι ένα μέγα τμήμα τη σημερινή ύφεση ε, οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας να ληφθούν γρήγορε αποφάσεις για την ολοκλήρωση, αποφάσεις που θα ενισχύσουν την Ευρωζώνη για την οικονομική διακυβέρνηση και για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στον πρόεδρο της Ευρωζώνης, το Eurogroup, τον κύριο Jean-Claude Juncker. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύον, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, με χαρά σας ξαναβρίσκω μετά από μια περίοδο διακοπών, που δεν ήταν ακριβώς περίοδος διακοπών, διότι αφιέρωσα περισσότερο χρόνο στο τηλέφωνο παρά στο τόπο τον οποίο ονειρευόμουν την περασμένη φορά που σας είδα. Ελπίζω η περίοδος δραστηριοτήτων η φετινή να είναι λιγότερο φορτωμένη από την περίοδο διακοπών που κανονικά θα είχα τον Αύγουστο. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω για να σας πω ότι όταν είχαμε την πρόθεση να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη στις αγορές γιατί αυτός είναι ο στόχος και το καθήκον ε, που έχουμε. Καλά θα κάναμε να εφαρμόσουμε τα όσα ε, ε, αποφασίστηκαν στις 21 Ιουλίου. Παρά κάθε μέρα να λανσάρουμε νέες ιδέες, αστόχαστα και καμιά φορά με τρόπο ανώριμο που δίνουν έδαφος για επιπόλες εκτιμήσεις και ερμηνείες ε, και εις βάρος των όσων τις κυκλοφορούν. Εγώ ε, πέρασα τις διακοπές μου στην Αυστρία, κοντά στη Βαβαρία, όπου έχουν ένα είδος μια παροιμία στη Βαβαρία που λέει ότι δεν θα πρέπει κάθε μέρα ε, να κυνηγάμε μια νέα ε, γουρούνα μέσα από το χωριό, να αμολάμε ένα γουρούνι και να το παίρνουμε από πίσω. Είναι μια παροιμία ε, αυτή η βαβαρέζικη, δεν ξέρω μεταφράζετε στις γλώσσες σας ε, και στο κόμμα σας παρακαλώ να το μεταφράσετε αυτό, όχι μόνο στη γλώσσα σας που είναι και δικό μου, αλλά ε, ελάχιστα, ελάχιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις 21 Ιουλίου και να μην βγάζουμε λαγό κάθε μέρα. Η στρατηγική των χωρών της Ευρωζώνης εγγράφεται στο πλαίσιο των αποφάσεων που είπαμε ελήφθησαν στις 21 Ιουλίου. Δηλαδή, θα πρέπει κάθε μέρα να ενισχύουμε σημαντικά τα μέσα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και μιλώ για το EFSF και το μελλοντικό μηχανισμό ε, σταθερότητας, για το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα και συμπαραμβανωμένο εδώ του τμήματος ε, που αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ε, για την εξυγίαση του ε, προϋπολογισμού και τη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας. Όλα αυτά θα αναφερθώ και τη διακυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αποφασίσαμε να λανσάρουμε ένα νέο πρόγραμμα μαζί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον ιδιωτικό τομέα εάν κατάφερε να εφαρμόσει η Ελλάδα το έκτακτο πραγματικά πρόγραμμα στο οποίο συμφωνήσαμε και οι τρεις. Δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή ότι η Ελλάδα θα είναι σε θέση να βγει από τη κατάσταση τη δύσκολη που βρίσκεται σήμερα. Τη στιγμή που σας μιλώ. Αποφασίσαμε, όπως είχα προαναγγείλει άλλωστε εδώ στην Επιτροπή σας, να μειώσουμε ε, τα επιτόκια δανεισμού για την Ελλάδα στο επίπεδο της διευκόλυσης, ε, δηλαδή περίπου στο 3% και μισό, 3,5%, όπως σας είχα προαναγγείλει εδώ, ε, με τη διάρκεια ε, των δανείων από 30 σε 15 χρόνια με μία δεκαετή περίοδο χάριτος. Αυτό που τότε ονομάσαμε profiling, ε, κάτι που οδήγησε σε σχόλια πάρα πολύ δυσάρεστα και ε, εις βάρος μου. Πάντως καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτή την επιμήκυνση. Το νέο ε, πρόγραμμα φτάνει στα 109 δισεκατομμύρια που έρχονται να προσταθούν στα 24 του προηγουμένου προγράμματος τα οποία ακόμα δεν έχουν εκταμιευτεί στο σύνολό τους. αυτά τα μέσα δεν θα καλύψουν μόνο τις δημοσιονομικές ανάγκες, αλλά θα βοηθήσουν να τονωθούν τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών σε μεγάλο βαθμό και θα βοηθήσουν ε, στην επαναγορά του χρέους. Και η Ελλάδα από μόνη της θα βελτιώσει τη ε, κατάσταση με τρόπο θεαματικό. Αυτό εξαρτάται από την τεχνογνωσία και από την επιμονή ε, της ε, ελληνικής κυβέρνησης στη δράση Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου θα δούμε την έκθεση της Τρόικα πριν μπορέσουμε να αποφασίσουμε για την εκτιδώση, την εκταμίευση συγκεκριμένα, που θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο. Γνωρίζετε ότι γίνεται μια συζήτηση τώρα για τις παράπλευρες εγγυήσεις ή απλώς εγγύησης για το ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα θέμα που έχει ανακοινήσει κυρίως η Φιλανδία και ακολουθώντας τη Φιλανδία ε, και άλλες χώρες ε, το ζήτησαν. Εμένα δεν μου αρέσουν ε, αυτοί οι μηχανισμοί, ούτε οι διμερείς συμφωνίες που γίνονται μεταξύ διαφόρων κρατών μελών. Γνωρίζουμε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Οι φινλανδικές αρχές και οι διαδοχικές κυβερνήσεις είχαν επιστήσει την προσοχή μας αυτό το φιλανδικό αίτημα που εντάσσεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Φιλανδίας, της νέας κυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, ε, υπεκφεύγει με ένα θολό τρόπο, σε μια όριστη διατύπωση και θεώρησαν οι δύο κυβερνήσεις ότι δικαιούνται να προχωρήσουν σε διμερή συμφωνία που με τον τρόπο που έγινε δεν ευσταθεί. Αναζητούμε τώρα άλλες λύσεις, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια λύση και δεν θεωρούμε ότι αυτό το θέμα των εγγυήσεων ε, θα μας εμποδίσει να μεταφέρουμε στην πράξη και στην πραγματικότητα ε, τις διάφορες αποφάσεις που ελήφθησαν στις 21 Ιουλίου, παράλληλα με τη σημερινή μας συνεδρίαση. Η ομάδα εργασίας ε, πραγματικά μελετά ε, τις ε, προτάσεις που πιστεύω θα ικανοποιήσουν όλα τα μέλη της Ευρωζώνης. Συμμετοχή τώρα του ιδιωτικού τομέα. Συνολικά εκτιμάται σε 135 δισεκατομμύρια ευρώ στα ομόλογα που λήγουν το 2011 από το 2011 μέχρι το 2020 και ανταλλάσσονται ε, με νέα μακράς διαρκείας. Η απώλεια ε, σε πραγματικές τιμές σημερινές θα είναι 21% για τον ιδιωτικό τομέα. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι γελή αυτή η απώλεια ή δεν είναι αρκετά μεγάλη. Πάντως σημειώνω ότι είναι σπάνιες εκείνες οι ευκαιρίες που ε, σε τέτοιες λύσεις τέτοιου τύπου. Είχαμε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα ε, αυτής της εμβέλειας. Δηλαδή το γεγονός ότι συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας και μόνο θα βοηθήσει να περιοριστεί κατά 12% το χρέος της Ελλάδας. Και αυτό αξίζει πραγματικά όλη μας την προσοχή και θα πρέπει να εκφραζόμαστε ε, ε, με τρόπο πιο επενετικό από ό,τι κάνουμε συνήθως. η ευελιξία του EFSF και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ε, θα ενισχυθεί σε τεχνικό επίπεδο. Την Παρασκευή το βράδυ βρήκαμε μια καλή απάντηση ε, στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και του πεδίου εφαρμογής ε, του Ευρωπαϊκού Προσωνού Μηχανισμού. Θα προσπαθήσουμε να λύσουμε κάποια τεχνικά προβλήματα τις επόμενες μέρες έχει επιτευχθεί συμφωνία για την αναθεώρηση ε, της συνθήκης που πρόσφατα υπεγράφει για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και βομένως ό,τι έχει σχέση με ε, τροποποίηση, μεταρρύθμιση του EFSF και ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ολοκληρώνεται αυτό τον καιρό. Μια συμφωνία που θα δώσει νέα πνοή. Για την Ιρλανδία θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από τις προόδους που έχει ε, επιτύχει. Η Ευρωζώνη Υποφέρει από το γεγονός ότι αβίαστα και καμιά φορά με χερεκακία διασπείρονται διάφορες αρνητικές ειδήσει και δυσάρεστες, ενώ τα θετικά δεν τονίζονται, δεν κυκλοφορούν. Η Ιρλανδία που ε, είχε ε, πολύ μεγάλες απώλειες ε, κατάφερε να τις καλύψει. Η Πορτογαλία, σε μεγάλο βαθμό, η Πορτογαλία που τώρα εφαρμόζει, αρχίζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα της, κάνει και αυτή μεγάλες πρόοδους και είμαι πολύ ικανοποιημένος από τα στοιχεία που ακούω από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που δεν μπορούν παρά να μας ικανοποιούν. Για την Ελλάδα είδομεν αφού λάβουμε γνώση ε, της έκθεσης της Τρόικα που αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα. Για την οικονομική διακυβέρνηση θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά επειδή είμαι σε 10 λεπτά και 27 ε, δεύτερα θα επιφυλαχθώ να απαντήσω και θα σας αφήσω τις εκπλήξεις για τις απαντήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Καταπληκτικό σας κοίταξα και αμέσως καταλάβατε. Φοβερό. Α ακούσουμε τον Επίτροπο Ρεν τώρα τελευταίο, αλλά όχι εξίσου σημαντικός με τους υπόλοιπου φυσικά. Σάρων, ευχαριστώ που με κοιτάζει έμονα. Uh, Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω στη σημερινή συνεδρίαση. Θα ήθελα να κάνω μια αποτίμηση των οικονομικών προοπτικών και της κατάστασης στις χρηματοπιστωτικέ αγορές. Μετά θα περάσω σε κάποια νομοθετικά ή μάλλον θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με την κρίση. Το καλοκαίρι εργαστήκαμε εντατικά σε συνεργασία με τον Jean-Claude όλος ιδιαιτέρως. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω σε μεγάλο βαθμό αυτά που σας είπε, κυρίως ε, για τα ζητήματα όπου συμφωνούμε. Για τα υπόλοιπα ε, θα δώσω την ευκαιρία στον Ζαν Κλώτ να συμφωνήσει μαζί μου μετά την ε, συζήτηση. In the first half of uh, this year. Κατά το πρώτο ήμιση του 2011 η ευρωπαϊκή οικονομία σταδιακά ανέκαμπτε βέβαια με ε, βραδύτερους ρυθμούς τώρα τελευταία. Παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ 0,8% το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο ε, ήταν βραδύτερη ανάπτυξη 0,2% και οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες ε, της ζώνης ευρώ υπέδειξαν ότι θα ε, ε, γίνουν τη βραδύτερη ρυθμή της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Έχουμε αυτά τα soft patches, τα επομονωμαζόμενα. Αυτή η βραδύτερη αναπτυξιακή ρυθμή δεν είναι ασυνήθιστη όταν μιλάμε για πολυετή προγράμματα ανάκαμψης και η ανάκαμψη αυτή έπεται μιας μεγάλης ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την δύσκολη κατάσταση και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Στις χρηματοπιστωτικές αγορές ε, ε, παρατηρείται μεγαλύτερη πίεση πλέον μετά το καλοκαίρι και φαίνεται ότι βιώνουμε μια παράλληλη επίδοση των χρηματοπιστωτικών αγορών ε, αφενός και αφετέρου της πραγματικής οικονομίας. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι. Πώς ερμηνεύω εγώ την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι χρηματοπιστωτικές ε, αγορές ε, και η ευρωπαϊκή οικονομία έχουν αρχίσει να συμβαδίζουν όλο ένα και περισσότερο ε, και έτσι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το spillover, την επιρροή των χρηματοπιστωτικών εξελίξεων επί της πραγματικής οικονομίας και κυρίως της απασχόλησης. Αυτό τονίζει το πόσο σημαντικό είναι να ε, περιορίσουμε τις χρηματοπιστωτικές διακυμάνσεις και έτσι να κατοχυρώσουμε την σταθερή οικονομική πορεία. Ε, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας έχουν επιδεινωθεί κατά τη σε σχέση με τις προβλέψεις που κάναμε την Άνοιξη και τώρα Εργαζόμαστε τις μεσοπρόθεσμες ε, προοπτικές ε, και θα τις κοινοποιήσουμε στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεδομένες της οικονομικής ε, και δημοσιοοικονομικής κατάστασης πρέπει να τονίσουμε την πολιτική απασχόληση. Σε ποιες επιλογές έχουν τα κράτη-μέλη για την μακροοικονομική τόνος δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα σε πολλά κράτη-μέλη δεν μπορούν να κάνουν τίποτα απολύτω. Άρα για να τονωθεί η ανάπτυξη χρειάζονται ε, ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, Έχουν λένε και πιο κέριο ρόλο δεδομένη της κατάσταση και πρέπει να ενταχθούν στη συνολική απάντηση που θα δώσουμε στην κρίση. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη λάβει σημαντικότατε αποφάσει τελευταίε εβδομάδε καθώς και μήνες κυρίως σε σχέση με τις ε, δημοσιοοικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις και άλλα διαρθρωτικά μέτρα που έχουν ε, βασικό αντίκτυπο ως προς την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Χρειάζονται ολένα και περισσότερα τέτοια μέτρα και επίσης για να είναι βιώσιμη η οικονομική μας ανάπτυξη ολένα και περισσότερο χρειάζεται να αναλάβουμε μέτρα χρηματοπιστωτικής διόρθωση. Ε, η κεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι σε μεγάλο βαθμό πολύ καλύτερη σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, παραδείγματο χάρη, και αυτό φάνηκε από τα στρες κοπόσεως που έγινε τον Ιούλιο. Οι ευρωπαϊκές ε, τράπεζες ε, αύξησαν κατά 50 δις ευρώ το μετοχικό τους κεφάλαιο ε, εν ώψη αυτών των τεστ και όταν κρίθηκε ότι ήταν αδύναμες οι κεφαλαικές θέσεις κάποιων τραπεζών μέσα από τα τεστ έπρεπε σε διάστημα 6 έως 9 μηνών να λάβουν μέτρα. Ε, σχετικά τώρα με τις ε, συγχωνεύσεις, την χρήση των ε, χρηματοπιστωτικών τίτλων λοιπά από τις τράπεζες προτείνονται κάποια μέτρα, αλλά προβλέπετε ότι όταν δεν υπάρχουν, δεν αναλαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα από τον ιδιωτικό τομέα, τότε θα πρέπει να παρέμβει ο δημόσιος τομέας. Παρόλα αυτά τα μέτρα ενίσχυσης της κεφαλαιοποίησης των ευρωπαϊκών τραπεζών παρατηρούνται δυσκολίες για την πρόσβαση ε, των τραπεζών ε, στις αγορές ε, τις τελευταίες εβδομάδες. Οι τράπεζες ε, αναμένουν οι όροι αναχρηματοδότηση να βελτιωθούν τις επόμενες εβδομάδες ε, και φυσικά οι τράπεζες έχουν πρόσβαση στην παροχή ρευστότητας από τις κεντρικές ε, εθνικές τράπεζες όπως ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο. Σε σχέση τώρα με τις αποφάσεις 21ης Ιουλίου, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ ανέπτυξε το θέμα εκτεταμένα. Εγώ θα ήθελα πριν κλείσω την παρέμβασή μου, να εστιάσω την προσοχή μου σε θέματα που σχετίζονται με την οικονομική διακυβέρνηση η ε, διαρκής αναζήτηση νέων ιδεών για να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Ε, είναι θετική, αλλά να μην ξεχνάμε τα όσα συνέβησαν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ε, την τροποποίηση των χρηματοπιστωτικών κανονισμών και την αρχιτεκτονική του συστήματος προληπτικής εποπτείας, καθώ και τους νέους μηχανισμούς EFSF και ESM. Το πιο σημαντικό όμω είναι το νομοθετικό πακέτο των έξι οδηγιών για την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό θα είναι βασικό θέμα, ε, βήμα συγγνώμη, για την ε, ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας ε, ώστε να καταστεί και πιο επίσημη η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ανισορροπιών παρατηρούνται μέσα στη ζώνη ευρώ. Γι' αυτό η έγκριση των έξι οδηγιών έχει ζωτική σημασία ούτως ώστε να μπορέσουμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόεδρο στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι η βασική νομοθετική βάση που χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω και να ενισχύσουμε και άλλα στοιχεία του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης. Η σύνοδο ε, του Ιουλίου κάλεσε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου σε στενή διαβούλευση με τον Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Eurogroup να εισηγηθεί συγκεκριμένα μέτρα μέχρι τον Οκτώβρη σχετικά με την αναβάθμιση του τρόπου λειτουργία και τη βελτίωση του μηχανισμού επίλυση κρίσεων μέσα στη ζώνη ευρώ. Ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να προσφέρουμε καλύτερη θεσμική διαφάνεια στη ζώνη ευρώ πέρα από την κοινοτική μέθοδο στήριξη. Ε, θα πρέπει συγκεκριμένα να δούμε πώς ακριβώς ε, θα χειριστούμε τις ε, ευθύνες ε, ανάμεσα στις, ε, ε, στη, στα συμβούλια ΕΚΟΦΗΝ και στα συμβούλια του Eurogroup επίσης πώς θα συντονίζουμε καλύτερα τις εργασίες ε, του Eurogroup, ποιες δομές θα χρησιμοποιούνται και ποιες θα είναι οι πρακτικές που θα ακολουθούνται για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων όλων αυτών των συνόδων. Επίσης έχουμε αυξημένες προσδοκίες σε σχέση με το μελλοντικό ενδυνάμει ρόλο των ευρωομολογιών ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση για το δημόσιο χρέος μέσα στην ζώνη ευρώ. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι ε, με όποια μορφή και αν εισαχθούν αυτά τα ευρωομόλογα θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από μια ουσιαστική και ενισχυμένη χρηματοπιστωτική εποπτεία καθώς ε, και συντονισμό των νομισματικών και οικονομικών πολιτικών ούτω ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω κινδύνους και να έχουμε πιο βιώσιμα δημόσια οικονομικά. Αυτό φυσικά θα έχει αναμφισβήτητα επιπτώσει ε, στην δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών και άρα απαιτεί μια έντονη συζήτηση στη ζώνη του ευρώ καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια συζήτηση λοιπόν για να διαπιστώσουμε αν ε, είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη να δεχτούν αυτό το σενάριο. Όπως είπα πριν από το καλοκαίρι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτής της δέσμης των έξι οδηγιών για την οικονομική διακυβέρνηση ανέλαβε δέσμευση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ταχύτερο μέλλον να εισηγηθεί μια εναλλακτική λύση για όλα αυτά τα τεχνικά ζητήματα για το σχεδιασμό ενό συστήματο ευρωομολόγων και επ' αυτή τη βάση και προτού κάνουμε οποιοδήποτε βήμα θα χρειαστεί ευρύτατη διαβούλευση για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν κοινοί παρονομαστέ και ποιο είναι ο πιο λογικό τρόπο να προχωρήσουμε. Ε, και ε, στον ε, στην επικείμενη ομιλία του ο πρόεδρος Μπαρόσο θα εκθέσει τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας με στη ζώνη ευρώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω στη συζήτηση που ακολουθεί στην παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τον κατάλογο των ομιλητών εδώ. Ας μην χάνουμε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πρώτος ο Ζαν Πολ Γκοζές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε ε, Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύον, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ καταρχάς που ήρθατε εδώ ενώπιόν μας σήμερα να μας μιλήσετε για την κρίση. δεν θα σας επικρίνω επειδή είστε παρόντες, εσείς είχατε το σθένος και το θάρρος να ερθείτε. Αλλά θα ήθελα να σας διαβιβάσω την αίσθηση πολλών βουλευτών. Μαθαίνουμε πολύ περισσότερα από τον τύπο παρά από τη θεσμική οδό. Και σήμερα είναι ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου. Μόλις μιλήσατε φεύγουν οι δημοσιογράφοι για να πάνε να διασπείρουν στα δίκτυα ε, τις ε, μικρές ε, φράσεις που κατάλαβαν να συλλάβουν να κατάφεραν να συλλάβουν. Δεν ξέρω ε, ίσως επειδή δεν έχουμε τις ίδιες ευθύνες, αλλά παρακολουθούμε τα πράγματα, αλλά υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Κάθε μέρα ακούν ε, συνεχώς στα ενημερωτικά δίκτυα οι πολίτες να γίνεται ο λόγος για την κρίση και διαβάζουν συνέχεια πρωτοσέλιδα. Και έρχονται και μας ρωτάνε, εσύ που είσαι ευρωβουλευτής, πες μας τι συμβαίνει. Και τι να του πω εγώ το καλοκαίρι, ότι διάβασα και εγώ όπως εσύ την εφημερίδα σήμερα το πρωί. Έγιναν ε, διάφορα πράγματα, αλλά είναι σημαντικό να πούμε ε, ότι υπάρχει και η κοινοτική μέθοδος και θα πρέπει να τη συζητάμε. Και θα ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε του ΕΚΟΦΗΝ ότι χαίρομαι για τα σταράτα σας λόγια για το τι πρέπει να γίνει ε, για το θέμα αυτό της διακυβέρνησης και την αντίστοιχη δέσμη. Ε, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, οι συνάδελφοι θα κάνουν ερωτήσεις και θα προτείνουν λύσεις. Δεν θέλω να μπω στα τεχνικά ζητήματα ότι τι μπορεί να κάνει κανεί όταν είναι βουλευτή. Αυτά που είπατε για το πακέτο της διακυβέρνηση όμω ε, έχουν σημασία. Αν θέλουμε να δώσουμε αξιοπιστία και στο Συμβούλιο αλλά και στο Κοινοβούλιο ταυτόχρονα θα πρέπει το σύντομότερο να καταλήξουμε για τη δέσμη αυτών των ε, θεμάτων. Δεν είναι τώρα ώρα να... Ε, αναλωνόμαστε σε λεπτομέρειες με σχολαστικό τρόπο κτλ. Ε, και ένα τελευταίο θα πρέπει να δείξουμε και στις αγορές, τις χρηματαγορές, όσο και αν δεν το θέλουν ορισμένοι, ότι υπάρχουν και όρια στην κλιμάκωση και στην κούρσα αυτή. Είναι χρήσιμα τα χρηματοοικονομικά για την πραγματική οικονομία, αλλά το καζίνο είναι επιβλαβές. Και η Ευρώπη, που δεν είναι μόνη της στον κόσμο, θα πρέπει να δείξει ότι υπάρχουν όρια στις απαιτήσει απόδοσης και αποτελεσμάτων. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, αν Ρωτήσετε τους αγρότες εάν είναι ικανοποιημένοι από τις επιδοτήσεις της ε, Ένωσης, θα σας πούν όχι. Το ίδιο ισχύει και με τα χρηματοοικονομικά. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε κάπου ένα όριο, ε, ε, μια ρύθμιση και για τα δημοσιοοικονομικά. Ενδεχομένως μέχρι να σταματήσουμε κάποιους κανόνες ε, να αποφασίσουμε ας πούμε, όπως είναι ο κανένας 11 ε, για θέματα ε, αφαιρικιότητας, χρεοκοπίας για να καθησυχάσουμε λίγο να καταγνάσουμε τα πνεύματα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος του Σοσιαλιστών Ούντο Μπούλμαν. Σας θυμίζω ότι έχουμε καθυστερήσει, γι' αυτό παρακαλώ να μείνετε στο χρόνο σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Γιούνκερ, κύριε Ρέν, ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον ότι ήταν σημαντικό για μας να ζητήσουμε και σωστό αυτή τη συνεδρίαση και ευχαριστώ ε, τις άλλες πολιτικές ομάδες που μας υποστήριξαν. Τώρα το θέμα είναι τι μήνυμα θα στείλουμε, τι θα πούμε. Τι μέλη γενέστε και τι θα πρέπει να ακολουθήσει τη σημερινή συζήτηση. Για μένα Δύο είναι τα βασικά σημεία. Πρώτον, αυτό φάνηκε από το φετινό καλοκαίρι, η μέθοδος της ε, διακυβερνητικής μικροσυνεννόησης δεν ε, ε, μπορεί πλέον να επιβιώσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα να βγούμε από την κρίση χωρίς να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει να δώσουμε στο Κοινοβούλιο ένα νέο χώρο. Τι σημαίνει. Είναι προφανές ότι όταν ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το EFSF, ε, ευθύς εξ αρχής έχει σχεδιαστεί, αν είχε μάλλον σχεδιαστεί και είχε εφαρμοστεί με βάση την κοινοτική μέθοδο, δεν θα είχαμε τις σημερινές δυσκολίες να κάνει μια χώρα διμερείς διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να θέλουμε ολίγη Ευρώπη. Παλαιότερα τα μεγάλα κράτη ε, συνεννοούνται για να αποφασίσουν για περισσότερη Ευρώπη και σήμερα συναντώνται για πολύ δευτερεύοντα ζητήματα. Και θέλω να ρωτήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου πότε ε, θα σταματήσει την πολιτική της εμπλοκή στο Συμβούλιο, πότε σκοπεύει στο θέμα ε, των ακάλυπτων ε, πωλήσεων του short selling για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να σταθεροποιήσουμε και τις χρηματαγορές. Σας ερωτώ και τους τρεις. Τα μηνύματα ε, της στασιμότητας, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιδράσουμε, γιατί είναι στασιμότητα. οι χρηματαγορές αντέδρασαν ε, στη συμφωνία για τον προπολογισμό στι ΗΠΑ και στη Γερμανία δεν προχωρούν τα πράγματα. Δηλαδή τι θα γίνει όταν λέμε για τι επενδύσει, τα λέει και η κυρία Λαγκάρτ, ε, που δεν είναι και καμιά ανόητη. Λοιπόν, ε, θα πρέπει να θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη κοινή Ευρώπη και όποιος δεν το επιθυμεί δεν πρόκειται να μας βγάλει από την κρίση. Μερικοί, ε, μερικές διμερείς περίπου σύνοδοι κορυφής δεν αρκούν. Ο κύριος Κλίντς από τους Φιλελευθέρους. Ευχαριστώ. Κύριοι και από πλευρά μου που ήρθατε ώρα μαζί να ε, συζητήσουμε, δείξατε αυτή την προθυμία. Ο Κίσιγκερ, πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, πάντα παραπονείται το ότι ποιο να πάρω τηλέφωνο στην Ευρώπη, ποιο είναι το τηλέφωνο της Ευρώπης, έχω τόσα τηλέφωνα. Και όταν πρόκειται για ε, τόσο σημαντικά θέματα και όταν ήθελε να συνεννοηθεί γρήγορα. Σε όλα αυτά τα θέματα που επίκυνται, για περαιτέρω συζήτηση. Έχουμε τον αρμόδιο επίτροπο, ε, τον προεδρεύοντα, τον πρόεδρο του Eurogroup, ε, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ε, σε λίγο θα έχουμε και ένα επικεφαλής της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό δεν βοηθάει για να δώσουμε την εμπιστοσύνη στους επικριτές και τους αρνητικούς ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αντί να απλοποιούμε τα πράγματα, τα περιπλέκουμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα κβαντικό άλμα, δηλαδή ο αρμόδιος επίτροπος να αποκτήσει περισσότερα δικαιώματα, όπως κάναμε για την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική. Γιατί δεν μπορεί ο αρμόδιος επίτροπος να ε, προεδρεύει, όπως λέει Άστον στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών, όπως κάνει εκείνη στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Γιατί δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερη ευθύνη και αρμοδιότητες ο αρμόδιο επίτροπο και να είναι προ τα έξω το πρόσωπο τη Ευρώπη ε, σε αυτά τα θέματα, για γυναίκα να είναι εκείνη η αρμόδια. Φοβούμε ότι με το δρόμο που έχουμε πάρει μέχρι τώρα δεν βελτιώνουμε την κατάσταση, παρά μόνο την επιπλέκουμε ακόμα περισσότερο και χρειάζεται ακόμα περισσότερες συνεννοήσεις και συμφωνίες σε μια κατάσταση που είναι έτσι και αλλιώς δύσκολη από αυτή τη σκοπιά. Ευχαριστώ. Η Κέιτ σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ όλου που ήρθατε σήμερα. Ο τίτλος της σημερινής συζήτηση είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών, νομοθετικές και θεσμικές απαντήσει. Οπότε στρέφομαι καταρχήν στην ανταπόκριση στη γνώμη των αγορών. Μετά από 18 μήνες, μετά από την αρχική ε, ελληνική κρίση χρέου. αυτή τη στιγμή φαίνεται να δίνουν 47% τα τριετή ε, ομόλογα, τα δεκαετή 14% και δεν μπορεί να γίνει κεφαλοποίηση για να αυξηθούν τα ε, χρήματα και η ΕΚΤ αγοράζει ερκώς από τη δευτερογενή αγορά. Άρα λοιπόν φαίνεται να μην εντυπωσιάζονται από τις απαντήσεις μας οι αγορές μέχρι στιγμής και υπάρχουν ε, τρεις τρόποι για να εξαλειφθούν ε, τα προβλήματα χρέους. Το πρώτο είναι το να εξαγοράσεις, το δεύτερο είναι το να μην το ξεπληρώσεις και το τρίτο είναι ε, να η υποτίμηση του νομίσματος. Η δεύτερη και τρίτη επιλογή δεν παίζουν, άρα ε, η σημερινή πολιτική πρέπει να είναι σαν να κάνουμε ε, ευχολόγιο για, να... για το μέλλον ε, η δική μας πολιτική αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα με τα προβλήματα που υπάρχουν και στην οικονομία της, των ΗΠΑ. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει σημαντική οικονομική ανάπτυξη, ποια είναι η εμπιστοσύνη σας ότι οι εθνικοί σας πολιτικοί θα μπορέσουν επιτέλους να ενεργήσουν αλτρουιστικά και να πείσουν την επενδυτική κοινότητα ότι το νέο πλάνο για την Ευρωζώνη μπορεί να λειτουργήσει συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων για την Ευρωζώνη και πέρα από αυτήν. Και Εφόσον υπάρξουν κονδύλια τα οποία θα προκύψουν από την ε, αγορά του, των χρεών, πώς θα μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση ώστε να αποφύγουμε την συνολική κατάρρευση. Και ευχαριστώ πολύ και εξ ονόματος του Πρασίνου ο κύριος Λάμπερτς. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους που είστε εδώ και περισσότερο ευχαριστώ γιατί περάσατε το μεγαλύτερο τμήμα του καλοκαιριού στην καταπολέμηση των πυρκαγιών. Θα πρέπει λοιπόν γι' αυτό και μόνο να σας ευγνωμονούμε, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με όλες τις αποφάσεις που λάβατε, πάντως σίγουρα δεν αφιστήκατε προσπαθειών. Καταρχήν να μιλήσω στον κύριο Γιούγκερ ως πρόεδρο του, του Ευρωγκρουπ για δύο θέματα. Όταν αρχίσουμε να διαβάζουμε με λεπτομέρειες τις υποθέσεις εργασίας και τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, μπορεί να υπάρξει, να διαπιστωθεί ότι μπορεί να είναι πολύ λιγότερο από το 21% επιπλέον, μια πολύ βασική εγγύηση για την αποζημίωση όλων των υπολείπων για την αποπληρωμή όλων των υπολείπων. Άρα λοιπόν αυτά για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα όπως αποκαλείται και να επανέλθω σε ένα σημαντικό σημείο, ένα από τα μέσα για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιας οικονομίας είναι βεβαίως ο τομέας των εσόδων. Και εδώ υπάρχουν και νούρια στοιχεία που προέκυψαν πριν και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πριν από το καλοκαίρι ήταν το γεγονός ότι η Κομισιόν σαφώς μας αποκάλυψε το πλωστάσιό τη όσον αφορά την εφαρμογή ενό φόρου για τις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και απευθύνομαι στο Ζαν Κλοντ και ως πρόεδρο του Ευρωγρούπου. Ποιες είναι οι πιθανότητες κατά τη γνώμη σας να μπορέσουμε όντω να καταλήξουμε κάπου με αυτή την ιδέα και να μετατραπεί σε πρόγραμμα βράχη πρόθεσμα, δηλαδή 2012-2013, τουλάχιστον στο πλαίσιο της, του Ευρωγκρούπ, αν όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Έπειτα, η συνεργασία του γαλλογερμανικού διδήμου μπορεί να σκεφτεί κανεί ότι θέλει αυτέ τι συνεδριάσει. Πάντω, ένα σημείο προσέλιξε την προσοχή μου, η ιδέα για πλήρη εναρμόνιση τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ε, ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Εσείς που το πώς τοποθετήσετε ως πρόεδρος του Ευρωγκρουπ, ξέρω πώς δεν είναι αυτός ο χώρος, αλλά εγώ θα ήθελα σίγουρα η Μπενελούξ να μπει σε αυτή την πρωτοβουλία αν τελικά πάρει μορφή. Οι οικονομίες μας είναι αλληλένδετες πλέον, πολύ συνδεδεμένες μεταξύ τους και γιατί όχι και φορολογική ένωση. Τώρα, για τα ευρωομόλογα συμμερίζομαι την ανάλυση του Όλη Ρεν. Είχε έτοιμη πρόταση. Είναι προφανέ ότι αν το φτιάξουμε αυτό, όχι μόνο θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον ε, εποπτεία, πρόκειται για ένα βήμα προ Ομοσπονδιακή Ευρώπη και εδώ χρειάζεται ευρύτερη συζήτηση, αλλά ξέρετε τουλάχιστον πω εμεί στηρίζουμε αυτήν την ιδέα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θαυμάζω ε, πάρα πολύ πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να μιλήσει γαλλικά. Ο κύριος Χοντής, παρακαλώ από την ΚΟΕ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια διαδικαστική πρόταση που έχει πολιτική ουσία. Συζητάμε σήμερα για τις οικονομικές εξελίξεις με τον Προεδρεύοντα, με τον Αρμόδιο Επίτροπο, με τον Πρόεδρο του Eurogroup. Δεν ξέρω πόσο ακόμα θα έχει αυτή την ιδιότητα και τους ευχαριστούμε πολύ που ήρθαν εδώ, αλλά νομίζω είναι προτιμότερο την επόμενη φορά, υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, να φωνάξουμε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή, γιατί όπως αποδείχτηκε, αυτοί λαμβάνουν αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακάμπτοντας τις συνθήκες και παρακάμπτοντας και τα θεσμικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεύτερο, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ύφεση που απειλεί όλη την Ευρώπη. Η παγκόσμια κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και είναι μπροστά μας και εδώ πρέπει να διαπιστώσετε κύριε Επίτροπε, κύριε Γιούνκερ, κύριε Προεδρεύοντα ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν για τη διαχείριση της κρίσης, νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αυτά τα προγράμματα λιτότητας στο όνομα των χαμηλών ελλημάτων και του χαμηλού πληθωρισμού είχαν σαν αποτέλεσμα να πλήξουν την πραγματική οικονομία, να θίξουν τους εργαζόμενους και να βυθίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ύφεση. Εδώ αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα κλπ. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της Ελλάδας. Πανηγυρίσατε ότι σώσατε την Ελλάδα με τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Έχετε πέσει έξω στις προβλέψεις. Μόλις πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Οικονομικών μιλάει για ύφεση 5% και όχι 3,8%. Η ανεργία φουντώνει, τα χρηματιστήρια βουλιάζουν, η υποειδιωτικοποίηση επιχειρήσεις έχουν χάσει το 30% της αξίας. Και εδώ σας ερωτώ κύριε Ρεν, σε ερώτηση που σας έκανα πριν λίγες μέρες γραπτή τι θα γίνει με τέτοιε τιμέ σημαίνει χάρισμα αυτών των επιχειρήσεων, μου απαντήσατε δώστε περισσότερε και σε γρηγορότερο διάστημα. Συμπέρασμα και θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Είναι δύσκολο κύριοι να είσαστε υπερέτε δύο σημεών, δύο αφεντάδων. Ή θα είσαστε εκπρόσωποι των συμφερόντων των λαών και των κρατών και τη υπόθεση Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα υπηρετείτε τι αγορέ. Και τα δύο δεν γίνεται. Επιμένω και επομένω και τελειώνω μήπως πρέπει επιτέλους να πάρετε κάποια μέτρα α, κερδοσκόπους, αγορές που τους χαϊδεύαμε τόσο καιρό που οδήγησαν σε αυτή την κρίση και που σήμερα βρισκόμαστε σε κρίση του τραπεζικού συστήματος όπως διαπιστώνει και η κυρία Λαγκάρτ να σταματήσει αυτό το χάιδεμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, αν συνεχίσετε όλοι να υπερβαίνετε το χρόνο σας, δεν θα καταφέρουν να μιλήσουν και οι τελευταίοι ε, ομιλητές στον κατάλογο. Να πω στον ε, Νικόλα ότι φυσικά υπάρχουν κάποιοι που θα απαντήσουν στο αίτημα αυτό να έρθουν ενώπιον της Επιτροπής, αλλά άλλοι σίγουρα δεν θα το δεχτούν. Ε? Η Μάρθα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε Ρεν είναι, φαίνεται μια θρησκεία πια, θρησκευτικό κανόνας, ότι οι οικονομικές αγορές είναι υπεύθυνε για την παγκόσμια κρίση και για την κρίση του χρέους. Η αντίδραση των αρχών, δηλαδή της Κομισιόν για τη ΣΕΣΜΑ, νωρίτερα αυτό το μήνα, όταν υπήρξε ανανεωμένη πίεση στις αγορές ήταν να αναζητήσουν ε, τις ακάλυπτες πωλήσει στην Ευρώπη. Φαίνεται ότι πρόκειται για τα μεγάλα οχυρά των ε, εμπόρων, αλλά μετά από την απαγόρευση των γαλλικών και των ιταλικών ε, τραπεζών, αυτές που προσπαθούσαν να προστατεύσει η Κομισιόν, από το που απαγορεύτηκε, λοιπόν πέσαν οι μετοχές αυτών των τραπεζών. Φαντάζομαι ότι οι μέτοχοι αυτών των τραπεζών δεν θα είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Ερώτημά μου προς εσάς είναι, θεωρείτε ότι η τράπεζα ε, ήταν επιτυχής για τις ε, μετοχές των γαλλικών και ιταλικών τραπεζών. Για τον κύριο Γιούνκερ, ε, σε σχέση με την επιδείνωση της κρίσης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, αυτό που σας προκάλεσε τα προβλήματα στις διακοπές σας και λαμβάνοντας υπόψη και το 17% των Ιρλανδών 70% συγγνώμη, του, των Ιρλανδών που δεν, δεν μπορούν να πληρώσουν τη δάνειά τους ε, και ζητούν βοήθεια. Τι θα κάνουμε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πλέον την κατάσταση και να επιτρέψουμε την κατάρρευση των ε, τραπεζών που δεν μπορούν να σταθούν και τις χώρες, χώρες οι οποίες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα να μην πληρώσουν τα χρέη τους. Ευχαριστώ. Ο Γκαρσία Μαργάλιο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Σάρων. Η πρώτη διαπίστωση σήμερα είναι ότι η αρχιτεκτονική δομή ε, όταν θεσπίσαμε το ευρώ που δημιουργήσαμε έχει αποτύχει. Θελήσαμε μια κεντρική νομισματική πολιτική, ένα κορσέ στις οικονομικές πολιτικές με μια υποτιθέμενη ανοιχτή μέθοδο συντονισμού δεν λειτουργήσε. Και τα υπόλοιπα τρία μέτρα, οι κανόνες που βασίζεται αυτή η αρχιτεκτονική έχουν καταρρεύσει. Το no bailout, το no default και ενδεχομένως αρχίζει να συζητείτε αν ε, θα αποτύχει και θα καταρρεύσει και ο κανόνας του no exit. Επίσης, το θέμα είναι της ε, λύσης της τραπεζικής κρίσης. Πριν από ένα χρόνο περίπου εγκρίναμε μερικές εκθέσεις ε, για την τραπεζική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά αργά και με βάση το τελευταίο προσχέδιο που ήρθα με λανθασμένο τρόπο. Δεν υιοθετεί τίποτα από όλα αυτά που είπε το Κοινοβούλιο. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Κατά την άποψή μου να αναγνωρίσουμε την αποτυχία ε, και να μην προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ε, την παλιά αρχιτεκτονική, αλλά να χτίσουμε μια νέα. Για τη δημοσιονομική πειθαρχία σας έχουμε πει ε, διάφορα θέματα από το Κοινοβούλιο, και να τα ακολουθήσετε. Για τα ευρωομόλογα και τα ε, ομόλογα λεγόμενα έργων, τα project bonds, για να έχουμε καλή διακυβέρνηση και να συνδέσουμε τη ε, δημοσιονομική πειθαρχία με ε, τα κίνητρα για την ανάπτυξη. Το Κοινοβούλιο επίσης έχει βάλει ένα πολύ συγκεκριμένο όριο ε, να μην μπορεί να μοιράζεται το χρέος αλλά τα ευρωομόλογα να συνδέονται με τη χρηστή και σωστή εφαρμογή των κανόνων. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη αρχιτεκτονική, πολύ καλύτερο σχέδιο, ευρύτερο, πληρέστερο και πιο μακροπρόθεσμο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Now... Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος Σοσιαλιστών ε, και Δημοκρατών Λεωνάρτο μπο... Ε, ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναπιστήσω την προσοχή σας σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και στρέφομαι πιο συγκεκριμένα στον, πρόεδρο, στον Επίτροπο Ρεν. Το πρόβλημα της βραδίτητας. Εγώ πιστεύω πως η ευρωπαϊκή πολιτική πάντα έρχεται μετά από τα γεγονότα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για αλλαγή ρυθμού από πλευρά της Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Και ρωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα είδος ε, think tank είναι όργανο διακυβέρνησης και πολιτικής κατεύθυνσης. Είναι σε, σε θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει σε, ενώπιον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, να έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκοντας έτσι ένα σύμμαχο για να προτείνει ένα πρόγραμμα μέσο και μακροπρόθεσμο με σαφή στόχου συγκεκριμένες προθεσμίες, με ένα είδος οδικού χάρτη που να μην είναι απλά επανάληψη των όσων γνωρίζουμε περισσότερο θάρρος και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Δεν μπορούν να δίνονται συνηθισμένες απαντήσεις σε έκτακτες καταστάσεις. Μία προοπτική ανάπτυξη ε, θα μπορούσε να αποτελέσει, ε, να δοθεί μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και η απάντηση στο πρόβλημα του χρέους ε, μπορεί να προέρθει μόνο από ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζονται νέα μέσα, γιατί διαφορετικά διερωτώ τι νόημα έχει η εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια ερώτηση ίσως λίγο αγαθή απευθυνθεί προς τον κύριο Γιούνκερ. Όταν γίνονται διασκέψεις κορυφής, γιατί στο τέλος κάθε μιας από αυτές δεν γίνεται προσπάθεια να εμπιστευθούμε σε μια επιτροπή, σε μια ομάδα εργασίας το την ε, αρμοδιότητα να προσφέρει μετά από τις διασκέψεις κορυφής μια αυθεντική ερμηνεία των συμπερασμάτων αυτής της διάσκεψης κορυφής και να εμπιστευτούμε μόνο σε αυτά τα συγκεκριμένα άτομα την αρμοδιότητα να μιλούν και να κάνουν ανακοινώσεις Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος του Έλκο Μάρκος Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, δύο ερωτήσεις. Ε, όταν συζητάμε ποιον θα καλέσουμε και τον κύριο Φαν Ρομπέ, αν ε, επιβληθεί αυτό που αποφάσισαν οι δύο στο Παρίσι. Και από την άλλη έχουμε και 17 εθνικά κοινοβούλια με τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους για την επικύρωση. Βλέπουμε με τρόμο τα τεκτενόμενα στη Φινλανδία. Ανα... αρχίσουμε να ζητάμε εγγύησεις για τα κρατικά δάνεια. Ε, καλή τύχη όταν συζητάμε ε, για άλλα θέματα και από ε, σαν αυτή που κατάγομαι εγώ. Είναι τελείως λαθασμένη αυτή η κατεύθυνση και η συζήτηση. Έχουμε ένα πρόβλημα δημοκρατίας τελικά. Κάποιες συμφωνίες ε, κυρίαρχων κρατών πώς μπορούν να γίνονται με τρόπο ε, που πρέπει να ε, επικυρώνονται από εθνικά κοινοβούλια. Εγώ για το ευρώ θεωρώ ότι τέσσερις πρέπει να αποφασίζουν. Ο αρμόδιος επίτροπος, ο, ο πρόεδρος του Eurogroup, αγαπητέ Ζαν ο πρόεδρο Κεντρική Τράπεζα, ο κύριο Βαν Ρομπέι, και άμα θέλετε κανέναν από το Συμβούλιο, α έρθει και εκείνο. Αυτή και στο δολάριο. Έτσι λειτουργεί και στην παλιά καλή εποχή πριν το ευρώ έτσι λειτουργούσε. Το λέω και στους ε, ε φίλους μου. Ε, ε, στη Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, την Bundesbank, εκατομμύρια ευρώ με τρία μηδενικά ε, επένδυε η Bundesbank για να σώσει το γαλλικό φράγκο, θυμηθείτε. Και άλλο ερώτημα, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, τι ρόλο διαδραματίζει εδώ σε αυτό το παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απαράδεκτο το θέμα του ευρώ να αφήνεται αποκλειστικά στα κράτη-μέλη και το θέμα της οικονομικής σύγκλησης, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι ε, πρόβλημα, να μην εξετάζεται και να μην το αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίσματα από τη Φινλανδία. <laughs> Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Φιλανδία. Ακούσα το Γερμανό συνάδελφο που δηλώνει ε, τρομοκρατημένο, ε, τρομοκρατημένος. Καταλαβαίνω γιατί. Γιατί εγώ εκλήθη να εξηγήσω στους ε, ψηφοφόρους μου γιατί η κυβέρνησή μας επιβάλλει αυτούς τους δυσάρεστους πολιτικά όρους. Αλλά πάντων το επεξεργαζόμαστε το θέμα προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι μεγάλο μέρος του κοινού πιστεύει πως ότι δεν φτιάξαμε το ευρώ για να είμαστε αλληλέγγυοι, το φτιάξαμε για κάποιους άλλους λόγους. Και έχουμε περιέλθει σε αυτή την κατάσταση όπου λείπει η εμπιστοσύνη και δεν υπάρχει ούτως ή άλλως αλληλεγγύη. Αυτή είναι η πολιτική κατάσταση που επικρατεί και επίσης ε, τι άλλο βιώνουμε η φινλανδική ε, Βουλή προσπαθεί να επιβάλλει όρους ε, που δεν μπορούν να δεχτούν άλλε κυβερνήσει. Τέλος πάντων αυτό πιστεύω εγώ, αλλά έχει διαφορετική άποψη το κοινοβούλιο μα. Άκουσα τα όσα είπε ο Ζαν Κλοντ σχετικά με αυτό το θέμα και περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω οι κύριοι ε, στο Προεδρείο τι πιστεύουν σχετικά με τι απαιτήσει της Φινλανδίας ε, γιατί φοβούμε ότι ε, είναι όλα αυτά κακή για το μέλλον ε, σχετικά με το συμπεφωνημένο πακέτο και το κάθε εξής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα που με απασχολεί. Μετά για το, τη δέσμη των έξι οδηγιών. Χαίρομαι που ο υπουργό Δροστόφσκι ε, έχει αναγάγει σε προτεραιότητα την εύρυθμη πορεία αυτής της δέσμης των έξι οδηγιών και είπε και ο Επίτροπος Ρέν ότι έχουμε καταφέρει ήδη πάρα πολλά, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να θυμηθούμε για ποιο λόγο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη το πακέτο, διότι κάποια κράτη-μέλη δεν προτίθενται να αναθεωρήσουν την πολιτική τους ή τις απόψεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Συμβουλίου και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα και πιστεύω πως πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι ένα θέμα αρχής και πρέπει με επικοδομητικό τρόπο να επιλύσουμε αυτό το θέμα που εκρεμεί. Προ το παρόν ε, ε, το Κοινοβούλιο εργάζεται με επικοδομητικό τρόπο και ευελπιστώ ότι θα βρεθεί μια λύση. Αλλά ε, εάν το Συμβούλιο δεν μετακινηθεί από τη θέση του, δεν υπάρχει λόγο αισιοδοξία. Αλλά ευελπιστώ ότι θα βρει, θέση το να, θα βρει μια λύση το Συμβούλιο. θα μπορούσαμε Επίση, να σχολιάσουμε τις ε, όχι και τόσο καλέ προτάσει σχετικά με το μέλλον της ε, οικονομικής ε, διακυβέρνηση, Ελπίζω όλοι να χρησιμοποιήσουν την ενέργειά τους για άλλα θέματα. Δεν ήσουν καλός Κάρλε, Ξεπέρασε το χρόνο σου από το ΕΛΚΑ. Ελπίζω να... Η κυρία Βόρτμαν Κόλ από το ΕΛΚ να είναι καλύτερη μαθήτρια και πιο πειθαρχημένη. Ευχαριστώ. Το ίδιο θέμα ήθελα να θέσω και εγώ με τον Γκάλ. Ως εισηγήτρια ε, θα ήθελα να τονίσω ε, και εγώ ότι θέλουμε να συμφωνήσουμε πάρα πολύ γρήγορα με το Συμβούλιο και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου για μένα υπήρξε κάποια ελπίδα, μια έκκληση να ολοκληρωθεί αυτή η νομοθετική προσπάθεια και ότι τα κράτη-μέλη θα υποστηρίξουν πλήρως την Πολωνική Προεδρία για να ε, συμφωνηθεί για την προληπτική δράση. Το ακούσαμε ε, σήμερα από τον πρόεδρο Τρισέ. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, ε, είναι πρόθυμο το Συμβούλιο να κάνει βήματα προς την πλευρά του Κοινοβουλίου. Και είναι ενδιαφέρον να ακούμε την επιβεβαίωση της Πολωνικής Προεδρίας και του Υπουργού Ροστόφσκη για τη θετική αυτή στάση ε, και την προθυμία να βρεθεί συμφωνία για το πακέτο αυτό το νομοθετικό. Η συνεχιζόμενη κρίση δημοσίου χρέου το καλοκαίρι μα κάνει να είμαστε ακόμα πιο πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα ψηφοφορία έτσι ώστε όλα τα κράτη να σέβονται τι δεσμεύσει του για τη δημοσιονομική τους πολιτική. Μικρά, μεγάλα κράτη είτε έχουν εκλογές του χρόνου είτε δεν έχουν ή αν τους λένε η Βλετέρμη η κυρία Μέρκελ, η κύριο Σαρκοζή. Όλοι θα πρέπει να εφαρμόζουν αυτά που τους αναλογούν. Χαιρόμαστε λοιπόν που το Συμβούλιο δέχτηκε αυτό το σύστημα αντιστραμμένης ε, ε, πλειοψηφία στη μακροοικονομική υποπτία, αλλά ο κρίκος που λείπει είναι ακριβώς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης να ε, εφαρμοστεί. Μπορούμε να αναμένουμε τις επόμενες εβδομάδες συγκεκριμένες κινήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, περιμένετε τις απαντήσεις στο τέλος. Υπερβάνους Περές από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να ξανακαλέσουμε τον Πρόεδρο Τρισέ ε, λόγω των ευθυνών που έχει για τα συστημικούς κινδύνους ε, και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Στιθερότητας γιατί αναρωτιόμαστε σε τι χρησιμεύουν αυτές οι προειδοποίησεις αφού τόσο ή άλλως ήρθε η κρίση και ήταν και καταστροφική όπως διαπιστώσαμε. Ε, Πρόεδρε Γιούνκερ είπατε δεν μου αρέσει αυτό που κάνει η Φινλανδία. Μα, μα γιατί μπόρεσε να το κάνει η Φινλανδία. Ούτε εσείς, ούτε ο Επίτροπος Δρέν, ο Πρόεδρος Μπαρός. γιατί δεν είπατε ότι όλα αυτά αντιβαίνουν πλήρως στο πνεύμα και στην ουσία της Συμφωνίας η Ιουλίου. Γιατί μετά την 21η Ιουλίου η κυρία Μέρκελ μπόρεσε να πει ότι ένα σχέδιο Μάρσαλ εγκρίθηκε για την Ελλάδα ενώ προφανέστατα ούτε οι αγορέ δεν το πίστεψαν ε, γιατί κατέρευσαν ε, οι αγορέ μετά την 21η και αυτό φυσικά δεν δείχνει ότι ανησυχούν για την έγκριση από τη πλευρά τη γαλλική κυβέρνηση και το Γαλλικό Κοινοβούλιο του Χρυσού Κανόνα δείχνουν αντίθετα την ανησυχία με τι προοπτικέ για τις επενδύσεις και για την ανάκαψη των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τώρα όμω που βλέπω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τη συνεισφορά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Σύνοδο τη 21 Ιουλίου ανησυχώ διότι ή μπορεί να μην ερμήνευσα σωστά τη δήλωση. Εγώ το, τουλάχιστον το μόνο που είδα είναι ότι ε, ε, μια προηγούμενη λύση σε σχέση με την Ελλάδα. Θα είμαστε λίγο πιο ελαστικοί σε σχέση με τους όρους εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτά διάβασα, μα συγγνώμη. Είναι αυτό σχέδιο ανάκαμψη, τόνο οικονομίας ή είναι σχέδιο Μάρσαλ. Θα ήθελα επίσης να θέσω άλλη μια ερώτηση. Η οικονομική διακυβέρνηση... Έχουμε αυτέ τι έξι οδηγίε, πολλοί σχολίασαν τη δέσμια αυτή και ασχολούμαστε όλοι με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι πιστεύετε με πάσα σοβαρότητα ότι μετά τι διακυμάνσει που είδαμε ε, τις τρικυμίες που είδαμε αυτό το καλοκαίρι μπορεί αυτό να αποτελέσει βάση συζήτησης, ε, δηλαδή το ευρωπαϊκό εξάμεινο επαρκεί και εν τη αυτή περίπτωση γιατί αφήνετε τον πρόεδρο Σαρκοζή και την καγκελάριο Μέρκελ να σχεδιάσουν τον οδικό χάρτη ενώ είναι δική σας η ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στην ερώτηση της Περβάς για το ρόλο του Τρισέ στον Πρόεδρο. Κανονικά έπρεπε να έρθει την Τετάρτη και ε, τον ε, φέραμε σήμερα. Δεν πρόκειται να μας ξεφύγει. Άλλη φορά θα ξανάρθει και θα απαντήσει ε, για το νομισματικό διάλογο. Τώρα, εξ ονόματος Λαϊκού Κόμματος, ο Βέρνερ Λάγκεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν αναλύσει κανείς Ποιες ήταν οι δυσκολίες στην αγορά. Κατά την άποψη μου ήταν η διαμάχη για τον προϋπολογισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, η υποβάθμιση της Αμερικής, ε, ε, δεύτερο, η τελείως άχρηστη επιστολή ε, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναστάτωσε τις αγορές και τρίτον η έγκριση των ειδικών συμφωνιών Ελλάδας-Φιλανδίας. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες ε, που μεσολάβησε το καλοκαίρι και του ίδιοι Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν συνεχίσουμε έτσι, οι χώρες που φέρουν ε, το μεγαλύτερο τμήμα των εγγύσεων δεν πρόκειται να συνεχίσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Σκεφτείτε και τις βουλές και τα κοινοβούλια των χωρών αυτών που καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνε στο ε, συνέχεια. Το είπε και η κυρία Βόρτμαν Κόλ προηγουμένω. Σαφώς, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, εμείς κάναμε μία προσφορά για το προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, σε μεγάλη ε, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Γιούγκερ που συμφωνεί, μπλοκάρουν η Γαλλία και η Γερμανία. Το μπαλάκι τώρα είναι σε εσά. Εσείς θα παραταχθείτε με την πλευρά του Κοινοβουλίου να δώσουμε αυτή τη μάχη εξουσίας. Η Γαλλία και η Γερμανία που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις και τις μεγαλόστομες ε, δεν είναι διατεθειμένες να υποχωρήσουν στα σημαντικά θέματα, δεν θα προχωρήσουμε. Και η τρίτη υπόθεση. Το καλοκαίρι ξεκίνησε μια συζήτηση για τα ευρωομόλογα. Κοινό χρέο μπορούμε να έχουμε μόνο αν αλλάξουμε τη συνθήκη. Αυτό είναι πρόγραμμα 2 και 3 ετών. Ενδεχομένως, αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, θα το σκεφτούμε τότε. Και δεν έχει νόημα να ορίσουμε μερικούς εκεί πέρα, αλλά μέσα στις συνθήκες να συμπεριληφθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με όλες τις υποχρεώσεις για να μπορεί να στέκει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά είναι τα θέματα και οι διαστάσεις που πρέπει να μας απασχολήσουν. Και όχι μια συζήτηση εξαμερικής ορμόμενη. Και εσείς πρόεδρε ανακατευθήκατε και ε, ε, κρίνεστε και ελέγχεστε χωρίς να έχετε ε, καμία δουλειά, καμία αρμοδιότητα, ούτε καν είστε μέλη της Ευρωζώνης. Και είπατε έτσι απότομα ότι δεν ήρθαν όλοι αυτοί που καλέσαμε. Μα οι τρεις που καλέσαμε ήρθαν και είναι και σωστοί. Πείτε το. Ποιον άλλον καλέσατε και δεν ήρθε, τον κύριο Μπαρόσο, ποιον άλλον. Δεν μπορείτε να το λέτε έτσι διαμία σε μια ερώτηση του συναδέλφου να καλέσουμε την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σαρκοζή και δεν ξέρω ποιον άλλον. Ξέρω εγώ και τον Πάπα. Και εσείς λέτε έτσι, εντάξει εμεί καλούμε κόσμο και δεν έρχεται. Ποιον καλέσατε παρακαλώ και δεν ήρθε. Uh, τον κύριο Βαν Ρόμπεϊ. Στο παρελθόν είχα καλέσει και τους Υπουργούς Οικονομικών της Γερμανίας και της Γαλλίας. Τελικά ήρθαν σε μια συνεδρία συντονιστών, αλλά σε ανοιχτή συνεδρία αρνήθηκαν να έρθουν ε, και έκανα μια γενική παρατήρηση. Μπορώ να καλέσω και άλλους, είμαι σίγουρη, αλλά ίσως θεωρήσουν ότι δεν είναι το σωστό πολιτικό επίπεδο για να έρθουν να απαντήσουν. Από πλευρά Σοσιαλιστών και Δημοκρατών τώρα, Τζιάννη Πιτέλα. Ευχαριστώ. Από πλευρά μου, πάρα πολύ ε, σύντομες ερωτήσεις, ε, σαν SMS. Πρώτο SMS. Ε, είναι ολιγορίες στην πολιτική και ε, ασθενής η πολιτική και αυτό βλάπτει. Η διακυβερνητική συνεργασία ε, με το πιο δύσκολο τρόπο και την πιο δύσκολη μορφή της. Η συνεννόηση του Διευθυντηρίου ε, Γερμανίας και Γαλλίας ε, έκανε ακόμα περισσότερη ζημιά. Πότε λοιπόν θα επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο SMS. Θα πρέπει το συντομότερο να βρούμε μια συμφωνία για τη διακυβέρνηση. Γεγονό είναι αυτό και σωστό. Αλλά επίσης θα πρέπει να επανισορροπήσουμε και τα κείμενα ή το κείμενο για την ανάπτυξη. Τους τελευταίους μήνες είδαμε ότι η ε, αναθεώρηση, μεταρρύθμιση της ε, διακυβέρνησης ε, μόνο στο σκέλος της δημοσιονομικής πειθαρχίας χωρίς ανάπτυξη ήταν ολέθρια. Τρίτο SMS, τα ευρωμόλογα. Δεν θέλουμε μια οποιοδήποτε λύση. Δεν είναι μια κάποια λύση. Είναι η μοναδική λύση για να βγούμε από την κρίση. Και εντάξει, μπορεί να το μελετάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ο ασθενή πεθαίνει. Πότε προτίθεστε να δράσετε. Ο πρόεδρος Μπαρόσο και εσείς ε, ο ίδιος ε, θα βοηθούσατε πολύ την Ευρώπη και θα ήσασταν πάρα πολύ χρήσιμοι ε, εάν λύνατε το χειρόφρενο. Οδηγείτε την Ευρώπη με το χειρόφρενο τραβηγμένο. Ε, πώς να προχωρήσει καμιά φορά μπορεί κανείς να αποφύγει ε, δυστυχήματα λύνοντας το χειρόφρενο. Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους. Δεν βλέπω την Πασκάλ εδώ πέρα. Σβέν, εσύ έτσι, από πλευρά των Πρασίνων. Μάλιστα. Θα ήθελα να θέσω κάποια ζητήματα. Πρώτον, για το θέμα των ευρωομολόγων. Δεν ήμουν σίγουρος ότι κατάλαβα καλά αυτά που λέγατε όλε. Εγώ ρώτησα το εξής. Θα δρομολογήσετε διαβούλευση. Ωραία, αλλά πρόταση θα κάνετε μετά. Είπατε ότι θα κάνετε τη διαβούλευση με όλους τους ε, συμμετέχοντες, ε, τους εμπλεκόμενους εταίρους, αλλά θα ε, επακολουθήσει και πρόταση. Η πρόταση θα είναι συνάρτηση του μοντέλου βέβαια και ίσως αυτό απαιτήσει περαιτέρω αλλαγές του μοντέλου οικονομικής διακυβέρνησης. Έτσι κατάλαβα τουλάχιστον. Όμως, άκουσα επίσης ότι, ε, από τους συναδέλφους ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένη πρόταση και γρήγορα για τα ευρωομόλογα. Δεύτερον, ε, διαπιστώνουμε τα προβλήματα ανάπτυξη ε, στην ευρωζώνη και ταυτόχρονα μειώνεται ο αριθμός των εναλλακτικών οδών και αυτό διαρκώς. Εάν κάποιοι δεν υποχωρήσουν και δεν παρετηθούν από κάποια από τα δικαιώματά τους, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στο μέλλον. Φυσικά ε, δεν αρκεί να λέμε ότι οι άλλοι πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές ελιτότητας ε, ταυτόχρονα. Θα πρέπει να δώσετε την ευκαιρία στο σύστημα να γνωρίσει την ανάπτυξη. Και αυτό δεν είναι Ζαν Κλοντ Ιουνκέρ ανέκαθεν ε, τα σώσουν υπέρ της μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Συμφωνώ και εγώ, αλλά τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή να προ... κάνεις μια εισήγηση για μια πραγματική ε, δημοσιοοικονομική ένωση. Το Λουξεμβούργο θα πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη, έστω και απίθανη πρόταση και ε, στο μέλλον να αδειμονώ να ακούσω τις προτάσεις σου. Θα είναι εξίσου επικριτικές και αυστηρές όπως τα σχόλιά σου για κάποιες χώρες. Ευχαριστούμε, αλλά υπερβαίνετε όλο το χρόνο σας από πλευράς ε, του ΕΛΚ. Εσάγια, ευχαριστώ. Όπως και ο συνάδελφος, θα παραδεχτώ και εγώ ότι είμαι από τη Φινλανδία. Όπως είπε ο κύριος Γιούνκερ στην ελακτήρια ομιλία του, μιλώντας για αυτή τη συμφωνία για τις εγγύησεις ε, που ζητάει η Φινλανδία. Ε, είπε λοιπόν ότι έγινε δεκτή η συμφωνία από όλες οι υπόλοιπες χώρες. Φαίνεται όμως τώρα ότι είναι ασαφή τα πράγματα. Όντως έγινε δεκτή. και εν τη αυτή περιπτώσει και άλλε χώρε θα ήθελαν αντίστοιχε ε, συμφωνίε όπω αυτή που έχει προγραμματίσει η Φινλανδία σε σχέση με την Ελλάδα. Ε, και είπατε ότι δεν απέχουμε πολύ από την εξέβρεση λύση ε, για αυτό το θέμα και θέλω να μου πείτε ακριβώ ποιε είναι οι υποσυζήτηση, η υποεξέταση λύση αυτή τη στιγμή, κάποιες έ έστω να μα δώσετε για τι περίφημε αυτέ λύσει. Κύριε Ρένε, θέλω να σα ρωτήσω το εξή Στη Φινλανδία έγινε μια πάρα πολύ έντονη εσωτερική συζήτηση. Αν ήταν δηλαδή σωστά ενημερωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την ε, ε, συμφωνία σε σχέση με τις ε, εγγυήσεις Φινλανδίας-Ελλάδας. Ήσασταν ενημερωμένος κύριε Ρέν και τι ακριβώς έγινε γιατί στην ε, Φινλανδία φαίνεται ότι θα οδηγηθεί σε ανατροπή η ίδια η κυβέρνηση λόγω αυτού. Οπότε μπορείτε να μας πείτε ακριβώς αν ενημερωθήκατε και ακριβώς γιατί ενημερωθήκατε ε, για αυτή την συμφωνία η Ιουλίου. Το σημαντικό στοιχείο ήταν η συγκατάθεση του ιδιωτικού τομέα σε σχέση με την μείωση των επιτοκίων δανεισμού και την παράταση ε, του χρόνου αποπληρωμής των δανείων φαίνεται πως ε, επικρατεί ασάφεια σε σχέση με το ε, πώς οι πιστωτές ε, προτίθενται να εφαρμόσουν αυτούς τους όρους. Μας δίνεται κάποια στατιστικά στοιχεία. Πόσες από αυτές τις τράπεζες συγκεκριμένα προτίθενται να υλοποιήσουν αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής από πλευράς των συντηρητικών είναι η Βίκη Φόρντ. Παρακαλώ πρέπει να τελειώσουμε στις και μισή. Οπότε ε, αν συμβαστεί το χρόνο σας θα ακούσετε και τις απαντήσεις. Βίκυ Φόρν. Ευχαριστώ. Στη δική μου χώρα δεν βλέπουμε μόνο πολύ μεγάλη αστάθεια στις αγορές, αλλά βλέπουμε και πολύ μεγάλη αστάθεια στους δρόμους. Και όταν βγαίνουν και αλληλοκατηγορούνται οι πολιτικοί, αυτό δεν βοήθησε ε, για να επανέλθει η ηρεμία, αλλά μόνο όταν οι κάτοικοι ε, των περιοχών αυτών υποστήριξαν ο ένας τον άλλον, μετά ε, οι τοπικές αρχές και μετά η πολιτική. Ε, αυτό είναι το δίδαγμα. Η πρόοδος δεν γίνεται όταν τα ρίχνουμε ο ένας τον άλλον και το φταίξιμο και τα λάθη, αλλά θα πρέπει να υποστηριχθούμε για να αντιμετωπίσουμε τις αγορές. Και βεβαίως και το ζήτημα του πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης είναι σημαντικό, αλλά σημαντικό είναι να έχουμε και ευθύνη, ε, γιατί είναι θέμα ε, κρατικού χρέους, δημόσιου χρέους και θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα για να βγούμε από αυτή την κατάσταση, για να επανέλθει ε, και η ευθύνη και η ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη φορολογία, αυτά που ακούστηκαν δεν νομίζω να βοηθούν ε, στην ανταγωνιστικότητα. Οι δοκιμές αντοχής της τράπεζας εντάξει ήταν πιο διαφανείς, καλά, αλλά ε, δεν ξέρω αν είναι ανταγωνιστικό. Το μοντέλο της βασιλείας ε, που επιτρέπει στις τράπεζες με μηδενικά κεφάλαια να επενδύουν στο δημόσιο χρέος νομίζω δεν ευσταθεί. Και πολλά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από κατάχρηση ε, αγοράς, από φήμες που δεν ευσταθούσαν ότι ορισμένοι θα ε, διώκοντο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τον πληθωρισμό. Το 2% ε, σου φαίνεται πολύ περισσότερο από 2% όταν δεν έχεις να φας, όταν δεν έχεις να βάλεις πετρέλαιο ή να κινηθείς. Γιατί ο κόσμος έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και ακόμα και το 2% είναι πληθωρισμός. Ευχαριστώ από το ΕΛΚ. Σλαβομίν Νίτρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα, συμφωνώ με τον κύριο Τρισέ και θα ήθελα να πω και εγώ στον Υπουργό ότι ε, μπορεί να έσωσε την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. θα πρέπει να δούμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Υπουργό, που είναι ακρεφνής υποστηρικτής της οικονομικής διακυβέρνησης. Πρόσφατα δηλώσατε στον τύπο ότι δεν διαχειριστήκαμε σωστά την κρίση. Αυτό πού το βρήκατε. Εισακουστήκατε στο Συμβούλιο από αυτά που είπατε. Ε, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και πώς μπορούμε να τα λύσουμε. Η Πολωνική Προεδρία τι θα κάνει ε, σε αυτά τα θέματα. Θα βοηθήσει να επιληθούν ή όχι. Έρχομαι τώρα στον κύριο Γιούνκερ. Ακούμε σήμερα πολλά και στεναρά και από τον κύριο Ρεν και από τον κύριο Ροστόφσκι ε, για ε, το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης. Εσείς κύριε Γιούγκερ συμφωνείτε, αυτό θα ήταν θετικό μήνυμα και προς τις αγορές. Συμφωνείτε με εκείνους που ε, ομιλούν υπέρ της νομοθετικής δέσμης. Είπατε κύριε Επίτροπε ότι ακόμα και όταν έχουμε περίοδο ανάπτυξης ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ε, μπορούν να έχουμε και περιόδους ε, μειωμένης ανάπτυξης, αλλά αυτό κινδυνεύει να ευρεωθεί. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Σίμων. Σήμερα συζητούμε για εμπιστοσύνη, για ηρεμία, αλλά αυτό που λείπει από τον κόσμο είναι η πίστη. Είδαμε το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, το πρώτο, και τι ζει η κοινή γνώμη. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην Ευρωζώνη ε, συμπεριφέρονται ε, σαν να κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις, προχωρούν, ε, φυγεί προς τα εμπρός, όλα τα λύσαμε, όλα εντάξει. Λίγο αργότερα έρχεται αυτό να ανατραπεί από κάποιους εξωτερικούς και να κλονιστεί η προηγούμενη απόφαση. Και τελικά ο κόσμος στην Ευρώπη δεν τα πιστεύει όλα αυτά. Όχι ο κόσμος στις χώρες που ε, ε, έχουν να κάνουν με προγράμματα ε, λιτότητας και μεταρρυθμίσεις, γιατί δεν βλέπουν φως στο τέλος του τούνελ, δεν βλέπουν μια προοπτική μετά από όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν το πιστεύουν ούτε εκείνοι που πρέπει να υπομισθούν την ευθύνη αυτή για τους ίδιους λόγους. Αν όμως τώρα από τον κύκλο των πολιτικών ακούγονται ε, αμφιβολίες και αν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους οι πολίτες μας, πώς θέλουμε να έχουν εμπιστοσύνη οι αγορές. Και κάτι που είπε προηγουμένως ο κύριος Μπούλμαν. Αυτό δεν, δεν θα γίνει με αλλαγή ε, της τακτικής, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αλλάξουμε τη μέθοδο με την οποία προχωρούμε. Δηλαδή χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη κοινοτική μέθοδος για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, αλλά και περισσότερη δημοκρατική συμμετοχή και δημοκρατικός έλεγχος απαιτείται. Άλλο σημείο αυτό. Επίσης, οι άνθρωποι στην Ευρώπη έχουν την αίσθηση ότι τους επιβάλλονται ε, αποφάσεις άνωθεν και δεν έχουν τρόπο να το επηρεάσουν παρά μόνο με ένα σταυρό που βάζουν σε ένα ψηφοδέλτιο στις ε, εθνικές εκλογές. Εδώ θα πρέπει να ζητήσουμε ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα και περισσότερη αποδοχή από την κοινή γνώμη, τον πληθυσμό της Ευρώπης και τελικά περισσότερη εμπιστοσύνη. Ζητώ συγγνώμη πρόεδρος, αλλά έχουμε φτάσει στο στάδιο που θα σας απαντήσουν μόνο στα αγγλικά γιατί θα μας φύγουν οι διερμηνείς. Από τους φιλελευθέρους το λόγο έχει ο κύριος Σκυλακάκης παρακαλώ. Ελπίζω να υπάρχει ακόμα διερμηνία. Η κρίση δεν αφορά μόνο στις ώρες χρέους. Στο μακροχρόνιο υπόβαθρο βρίσκεται και η διαφορά μεταξύ των ρυθμών βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωζώνης, κυρίως μεταξύ Βορρά και Νότου. Η σημερινή απάντηση στο πρόβλημα ο αποπληθωρισμός είναι εφιαλτικά δύσκολη για τα περισσότερα πολιτικά συστήματα. Οι αυτόματες κυρώσεις θεωρητικά θα λύσουν το πρόβλημα της ισόρευσης νέων ελλημάτων. Ποια όμως είναι η απάντηση της Ευρωζώνης στη συσσόρευση νέων διαφορών στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας τη καινοτομία, που σίγουρα θα έρθει στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει απάντηση χωρίς πολύ βαθύτερη και με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα ευρωπαϊκή ενοποίηση. Και δεν αναφέρουμε εδώ σε κάποια νέα στρατηγική της Λισαβόνας ή τέτοιου είδου αποτελεσματικότητα πολιτική. Και δύο σύντομε ερωτήσει στον Επίτροπο Ρεν που αφορούν την κρίσιμη για όλου μας πορεία του ελληνικού προγράμματος εξυγίανση. Μίλησε και συνάδελφο Άλλο Τι επίπτωση θα έχει η βαθύτερη της προβλεπόμενης ύφεση που ανακοινώθηκε πριν μερικές μέρες από τις ελληνικές αρχές στους δημοσιονομικούς στόχους για το 2011. Είναι πολύ κρίσιμη η ερώτηση αυτή για την Ελλάδα. Και η δεύτερη, τα στοιχεία δείχνουν ξανά και ξανά ότι η έμφαση στην αύξηση της φορολογίας, στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα κατά 50%, δεν φέρνει τα αναμενόμενα έσοδα με δεδομένη την ύφεση και την ποιότητα του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Πώς τελικά θα επιτευχθούν οι στόχοι, με στροφή στην περικοπή δαπανών και στην ταχύτερη υλοποίηση των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων ή θεωρεί ο Επίτροπος ρεαλιστική την επίτευξη των στόχων μέσω νέας φορολογίας. Σας ευχαριστώ. Σα e Σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος ε, του Έλκη Ντανούτα Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την Πολωνική Προεδρία για την ανάπτυξη. Γιατί η Πολωνική Προεδρία έθεσε την, ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολωνική κυβέρνηση ε, είχε, ήταν επιτυχής στο να βρει το σωστό μείγμα πολιτικής ώστε η οικονομία πραγματικά να αναπτυχθεί. Και είναι αλήθεια πως ε, η Ευρώπη χρειάζεται ε, ανάπτυξη. Δεν είμαστε σε αυτό διχασμένοι. Οι πολιτικοί, οι θύνοντες όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται τις διαρθωτικές ώστε να υπάρξει αντίκτυπος στην ανάπτυξη. Όμως είμαστε διχασμένοι όσον αφορά την μακροοικονομική πολιτική και το μείγμα αυτής που χρειάζεται ώστε να υπάρχει χώρος ε, για την Ευρώπη για να αναπτυχθεί και είναι γεγονός σήμερα ότι παρακολουθούμε ένα παράξενο μονοπάτι περιοριστικής νομισματική πολιτικής και ψηλότερη φορολογία. Και αυτό φυσικά δεν αφήνει περιθώριο για ανάπτυξη. Αν δούμε λοιπόν πώς αντιδρούν οι αγορές ομολόγων ιδιαίτερα, δεν ενδιαφέρονται μόνο για το χρέη, αλλά και για το δυναμικό ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Άρα λοιπόν το σχόλιο μου είναι πώς βλέπετε τη μελλοντική πολιτική και Ειδικά όταν ακούμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα συνεχιστεί αυτή, αυτό το μονοπάτι της περιοριστικής ε, πολιτικής, πώς θα αποφύγουμε επανάληψη αυτού που ζήσαμε το 2008. Ε, Σας ευχαριστώ και τώρα ο Ενρίκε Σαλόν. Ευχαριστώ. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν στο δύσκολο καλοκαίρι που περάσαμε και η συντρόφισσα υπερβάς ε, ιδιαίτερα μίλησε για ολέθριο. Αλλά μήπως είναι τώρα πιο θερμό το φθινόπωρο και πιο δύσκολος ο χειμώνας. Γιατί έχουμε τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος και του χρέους και έρχεται να προσθεθεί τώρα και ανησυχία σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξη. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος τώρα είναι η ανάπτυξη. Το είπε και ο Τρισέκ και ο κύριος Όλη Ρέν ότι είναι χαμηλή η ανάπτυξη, έστω και αν υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική πολιτική με ενθάρρυνση, με κίνητρα για την ανάπτυξη. Αυτό ανέκαθεν το έλεγε η πολιτική μας ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και γνωστοί κάτοχοι βραβείου Νόμπελ και τώρα έρχεται να το υιοθετήσει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική για την ανάπτυξη. Η χώρα μου, η Ισπανία, λαμβάνει αποφάσεις τώρα για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη. Ε, ε, συνταγματική αναθεώρηση με ευελιξία, νομοθετικές εξελίξεις και μεγάλες πολιτικές συμφωνίες. Αλλά ε, θέλουμε και πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη δεν θα πρέπει να είναι μόνο στα δημοσιονομικά αλλά και στα θέματα της ανάπτυξης. Γι' αυτό ερωτώ ε, και τους τρεις ε, προσκεκλημένους τι σχέδια έχετε για να τονωθεί η ανάπτυξη. Και τέλος άκουσα μια παρέμβαση που έλεγε ότι το ευρώ δεν δημιουργήθηκε για την αλληλεγγύη. Και πρέπει να τονίσω ότι το ευρώ δεν είναι σκοπός, είναι μέσον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ένωση όμως μεταξύ των αξιών και των βασικών στόχων έχει την αλληλεγγύη. Και θα πρέπει να πω ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο οικονομική. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές όπου πάρα πολλές χώρες δείχνουν αλληλεγγύη με τις υπόλοιπες. Thank ευχαριστώ πολύ και μια τελευταία σύντομη ερώτηση από τον Μάριο Μάουρο. Σα ευχαριστώ. Ωραία ήταν αυτή η μετάφραση της βαβαρικής ε, παροιμίας. <laughs> Αλλά πρέπει να μου εξηγήσετε και τι σημαίνει. Να ρωτήσω λοιπόν εγώ τον πρόεδρο Γιούνκερ τι πιστεύει με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει για τα ευρωμόλογα. Και το λέω γιατί όταν, πήρατε, όταν μιλήσατε τις περασμένες, μίλησε μάλλον τις περασμένες μέρες, ο πρόεδρος Φαν Ρομπαϊ πάγωσε τις προσδοκίες γιατί είπε ότι λείπουν ε, τα στοιχεία συνένεσης για να κινηθούμε προς τα ευρωομόλογα. Σας ρωτώ λοιπόν, χωρίς να περιμένουμε αυτές τις μελέτες και κόντρα μελέτες της Επιτροπής, ποια είναι αυτά τα στοιχεία συνένεσης, τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσει για να ανοίξει ο δρόμος για τα ευρωομόλογα και ως προς αυτό κάθε κυβέρνηση να κινηθεί ώστε να θέσει σε, σε ψηφοφορία τους ισολογισμούς. Μπορεί αυτό να, να ανοίξει το δρόμο για τα ευρωμόλογα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ συνάδελφοι που με ανεχτήκατε γιατί ήμουν λίγο πιο αυστηρή. Νομίζω ότι θα ακούσουμε με την ίδια σειρά όπως και στην αρχή τους ε, ομιλητές. Καταρχήν να ρωτήσω τον κύριο Ροστόφσκι να πατήσει. Ε, αν μπορείτε να μιλήσετε για 8 λεπτά, ίσως και αν τα καταφέρουμε μέχρι τις 6.30. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό που είπατε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε όχι για την αλληλεγγύη αλλά για κάτι άλλο ίσως να είναι αλήθεια. Αλλά αν δεν ε, επιδείξουμε την αλληλεγγύη που χρειάζεται για να σωθεί το ευρώ, τότε όλα τα υπόλοιπα πράγματα για τα οποία δημιουργήθηκε το ευρώ, δηλαδή μια αληθινή εσωτερική αγορά, ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη, μεγαλύτερη ευημερία για τους λαούς μας, τότε βέβαια θα είμαστε σε πολύ δυνότερη θέση από ότι αν δεν, αν, δεν είχαμε καθόλου φτιάξει το ευρώ καταρχήν. Και νομίζω πως αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη Βόρεια Ευρώπη. Ότι δηλαδή ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί πως ακόμα και αν κάποιοι πιστεύουν πως η δημιουργία του ευρώ ήταν λάθος, δεν είναι και κάτι από το οποίο μπορούν να ξεφύγουν χωρίς συνέπειες. Πολύ βαθιές συνέπειες μάλιστα. Mm. Η Κέιτ Winburn είπε ε, ότι, οι αγορές δεν έχουν πιστεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε πείσει εμείς. Εμείς δεν πείσαμε τις αγοράς. Δεν τα καταφέραμε. Και βεβαίως Αυτά τα λέω χωρίς ε, φυσικά καμία απολύτως ικανοποίηση. Και ως Πολωνός υπουργό Οικονομικών, του οποίου η χώρα δεν είναι στην Ευρωζώνη, εγώ μπορώ μόνο να μιλήσω για τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει αυτή η αποτυχία, για αυτό που ίσως θα θέλαμε να αποκαλέσουμε αθώου ε, παρατηρητέ. Θα έχει λοιπόν τεράστιες συνέπειε και πιστεύω ότι θα είναι εξίσου μεγάλες οι συνέπειες και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και γι' αυτό ο Τζος και εγώ λέμε πως ε, ανέκαθεν ήμασταν υπέρ της βαθιάς ολοκλήρωσης, την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την Ευρωζώνη, ώστε αυτή να διατηρήσει τη σταθερότητά της για την ε, δέσμη των έξι οδηγιών. Ε, ναι, θα εργαστούμε εντατικά με την συμφωνία των κυβερνήσεων ώστε να βρεθεί μια λύση όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν πρόκειται να αφιστούμε προσπαθειών δεν θα λείψουμε από καμία συνάντηση που θα μας δώσει μια ευκαιρία για να πετύχουμε γρήγορη ολοκλήρωση της υπόθεσης αυτής. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω ότι είναι ζωτική σημασία στο να κινηθούμε γρήγορα Και μάλιστα δεν μπορώ να το πω αυτό χωρίς να είμαι έτοιμος εγώ να παίξω πλήρως τον ρόλο μου. Και το λέω αυτό έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών μου. Ότι θα κάνουμε δηλαδή ό,τι μπορούμε ως Προεδρία για να εξασφαλίσουμε την εξέβρεση συμβαστικής λύσης. Και νομίζω πως αυτό απαντά και σε άλλες ερωτήσεις. Για την ανάπτυξη είδαμε πέρυσι μια σημαντική αλλαγή διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιστεύουμε πλέον ότι η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα ωραίων πραγμάτων όπως ε, οι δαπάνες στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Διαπιστώνουμε πως η ανάπτυξη είναι ε, συνέπεια δυσάρεστων πραγμάτων όπως η απελευθέρωση των ελεγορών εργασίας, η αφαίρεση των διάφορων εμποδίων και ακάμπτων σημείων και είναι πλέον ε, η κατάλληλη στιγμή για να διαπιστώσουμε πως οι διευθυντικές αλλαγές δεν είναι μόνο για τις αναδυόμενες αγορές, αλλά ίσως και κυρίως και πρωταρχικά για την Ευρώπη. Για το θέμα της διαχείρισης της ε, δημοσιονομικής πολιτικής, Είμαστε κοντά στα όρια της δημοσιονομικής πολιτικής, μάλλον στο εύρος της ε, δημοσιονομικής πολιτικής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένων και των μεγαλύτερων, ορισμένων μάλλον εκ των μεγαλύτερων και γι' αυτό Συμφωνώ με την Ντανούτα Χούμπνερ ότι αν η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να δώσει κίνητρα, τότε η νομισματική πολιτική θα πρέπει να προσαρμοστεί στην κατάσταση. Δεν συμφωνώ μαζί της ότι η Κεντρική Τράπεζα λέει πως ε, θα προχωρήσει στην φάση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής σε αυτό το μονοπάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω έτσι τα λόγια της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά έχουμε ένα βασικό πρόβλημα ότι δηλαδή κάποια από τους προϋπολογισμούς μας, κάποια από τις οικονομίες μας είναι υπό τεράστια πίεση και δεν θα ήταν λογικό να υπάρξει μια κατάσταση κατά την οποία όλοι δεχόμαστε πως ορισμένε ε, τράπεζες είναι εξαιρετικά μεγάλες και δεν επιτρέπεται να καταρρεύσουν, αλλά φαίνεται να δεχόμαστε ότι τις μέρες οικονομίες είναι αρκετά μικρές ώστε να καταρρεύσουν. Όχι, καμιά οικονομία δεν είναι αρκετά μικρή ώστε να τις επιτρέψουμε να αποτύχει και να καταρρεύσει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και η ΕΚΤ κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όλοι αισθανόμαστε σαν να θέλουμε να χειροκροτήσουμε, αλλά να προχωρήσουμε στον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Κυρία Πρόεδρε, κάποια σύντομα σχόλια, έτσι καταληκτικά. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι οι χρηματαγορές δεν επίστησαν ε, από τα όσα πράξαμε, είναι γεγονός αυτό, δεν επίστησαν. Διότι δεν ε, είμαστε και άριστοι στην επικοινωνία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ε, ούτε μένα με πείθουν οι χρηματαγορές. Έχω μείνει άναυδος μπροστά σε αυτή την αφέλεια του πολιτικού κόσμου. Ε, με έτσι οικουμενική εκπροσώπηση που θεωρεί ότι οι χρηματαγορές έχουν πάντα δίκιο και εμείς έχουμε πάντα άδικο. Μα πού βρισκόμαστε επιτέλους. Αυτοί οι ίδιοι που ζητούν την κυριαρχία της πολιτικής στις χρηματαγορές είναι οι πρώτοι που επικρίνουν εκείνους που απευθύνονται στις χρηματαγορές με τρόπο που δεν τους αρέσει των χρηματαγορών. Ο πολιτικός κόσμος υπάρχει για να ε, είναι το παπαγαλάκι των χρηματαγορών αυτό είναι ο διάλογο μας με τις χρηματαγορές, να επαναλαμβάνουμε το όσα μας λέγουν. Έχουμε συμφέροντα να υπερασπίσουμε. Και πώς θέλετε. Εγώ δεν βάζω αυτό σε εξίσωση. Δεν εξισώνω τις χρηματαγορές, δεν τι ταυτίζω με τους κερδοσκόπους. Αλλά πώς θέλετε να πείσετε τους κερδοσκόπους. Δεν πρόκειται ποτέ να πεισούν οι κερδοσκόποι. Όταν όμω απευθυνόμαστε στι χρηματαγορές, θα πρέπει να του μιλάμε ως ε, υπεύθυνοι πολιτικοί. Εμείς είμαστε στην υπηρεσία των λαών μας και όχι στην υπηρεσία των χρηματαγορών. Οπότε θα πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να αντιμιλούμε και στις χρηματαγορές και να τους εναντιονόμαστε και να μην ε, απορούμε κάθε φορά και ε, ε, όταν βλέπουμε κάποιο πολιτικό να αντιτίθεται στις χρηματαγορές. Σε ό,τι αφορά το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών δεν είναι πρόσφατη επινόηση γαλλογερμανική. Εδώ και καιρό υπάρχει στα κείμενά μας θα έλεγα βεβαίω. είμαι ε, πολύ υπέρ αυτή τη προσπάθεια, ε, αν μη τι άλλο και για λόγους δικαιοσύνη και καλύτερης αποδοχής ε, από τους λαούς της Ευρώπης των όσο κάνουμε στην Ευρώπη. Θα ήθελα όμως αυτό να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν πρόκειται. Οπότε, ε, δεν θα επιμείνω πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα να γίνει σε επίπεδο 27, επίσης δεν πρόκειται, οπότε δεν θα επιμείνω. Ε, τότε θα ήθελα να γίνει σε επίπεδο ε, Eurogroup. Εγώ, Juncker, μιλάω προσωπικά και όχι εξ ονόματος του Eurogroup. Γιατί θεωρώ ότι ε, αν δεν αρχίσουμε από κάπου να δίνουμε το παράδειγμα στον πλανήτη, δεν πρόκειται ποτέ να μας ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Και το λέω έχοντας υπόψη μου τις κακές εμπειρίες της Σουηδίας. Προσωπικά όμως είμαι υπέρ μιας τέτοιας προσέγγιση σε επίπεδο Eurogroup. Είμαι και υπέρ της ε, ε, Δημοσιονομικής Ένωσης. αυτό μας έλειπε, να έρθουν οι πράσινοι να μας το εξηγήσουν. Όσοι γνωρίζουν, δεν είναι πολλοί, αλλά γνωρίζουν, θα πρέπει να εξηγήσουν την περίεργη κατάσταση και σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη δημοσιονομική πολιτική και το Λουξεμβούργο. Δύο ώρες σκοτωνόμουν να εξηγήσω ε, αυτή την ερωτική σχέση, αυτό το ιδίλιο που υπήρχε ανάμεσα σε εμάς και στη Δημοσιονομική Ένωση. Αλλά κάθε φορά που έγινε πρόοδο στην Ευρώπη, δημοσιονομική, ε, κάθε φορά που γινόταν ε, και φορολογική ήταν σε Λουξεμβουριανή Προεδρία. Ε, ΦΠΑ, ειδική φορή κατανάλωσης, ε, ε, φόρος ακίνητης περιουσίας. Σταματήστε αυτό το παιχνιδάκι ή καλέστε με στην ομάδα σας. Μην με κάνετε να χάνω το χρόνο μου κάθε φορά στην Επιτροπή για να σας τα λέω αυτά τα φορολογικά και οι σχέσεις Λουξεμβούργου φορολογίας. Το Δεκέμβριο του 1997 βεβαίως πάλι στην Προεδρία του Λουξεμβούργου ή στην περίπτωση του συντονισμού των μεγάλων μακροοικονομικών πολιτικών μας θα κοπανάτε συνέχεια αυτά ε, για τη φορολογία. Διαβάστε το αυτό παρακαλώ προσεκτικά, μελετήστε το και θα μάθετε πολλά από τα κείμενα τα οποία δημοσιεύτηκαν για να ξεχαστούν στη συνέχεια. Και επίσης θα διαπιστώσετε, σημειώσετε ότι δεν νοείται φορολογική ένωση χωρίς ε, κοινωνική ένωση. Γιατί να έχουμε παντού την ίδια φορολογία αν δεν έχουμε ελάχιστο κοινωνικό μισθό, κατώτατο μισθό στην Ευρώπη για να έχουμε και ελάχιστους κανόνες ε, στις απολύσεις και ελάχιστου κανόνες στα δικαιώματα των εργαζομένων. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να ζητάω ελάχιστα δικαιώματα ανέκαθεν κοινωνικά για τους εργαζομένους. Το έλεγε και ο Ντεγκόλ. Ότι είναι τεράστιο πρόγραμμα, αλλά ο Ντεγκόλ ήταν ο Ντεγκόλ. Αυτό να δείτε πόσο τεράστιο πρόγραμμα και ο Ανός είναι. Σε ό,τι αφορά τις εγγύσεις που ζητάει η Φιλανδία, στη ε, συνεδρία στο Eurogroup, ο, όλοι και εγώ, ποτέ δεν υποστηρίξαμε αυτό το αίτημα, την αξίωση της Φιλανδίας. Προσπαθούσαμε να το κατανοήσουμε. Το Συμβούλιο έκανε μια αόριστη διατύπωση ε, για να συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μετά έρχονται και μα ζητάνε τα ρέστα στο Eurogroup και να το λύσουμε το πρόβλημα. Θα το κάνουμε. Και δεν θα σας πω κυρία μου πώς, διότι ε, είναι καθοδόν ακόμα οι διαπραγματεύσεις, αν το έλεγα τώρα, προφανώς η λύση δεν θα βρισκόταν ποτέ. Προσπαθώ να σιωπήσω. Έχω όμως κάποια ιδέα για ορισμένα θέματα. Σε ό,τι αφορά τη δέσμη των έξι οδηγιών, σε όσους με ρωτούν, απαντώ ότι, δεν σας λέω τίποτα καινούριο, ε, απαντώντας ότι εγγράφομαι πλήρως στη γραμμή του Κοινοβουλίου. Η εισηγήτρια το ξέρει πολύ καλά και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Eurogroup παντού λέγω ότι και εγώ και οι δύο άλλες κυβερνήσεις του Μπενελούξ είμαστε μαζί με το Κοινοβούλιο. Ε, γιατί με καλείτε να επαναλάβω ε, όσα έχω πει. Έχω πλήρη πιστοσύνη στο Γιάτσεκ ότι θα προχωρήσει. 21 Ιουλίου διήκρινα ε, κάποιες ε, πρόοδους ε, από γειτονικά κράτη, από κάτι δημοκρατίες γαλλόφωνες, ότι ορίστε ας το αποφασίσουμε τώρα. Δεν το αποφασίσαμε στις 16 Ιουλίου, θα το αποφασίσουμε τώρα. Πάντα αφήνουμε τα πράγματα να χρονίζουν και τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις και τις χρηματαγορές. Ενώ έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας για να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις στην κατάλληλη και σωστή χρονική στιγμή. Είμαι λοιπόν ε, ε, στο πλευρό του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση. Τίποτα καινούριο δεν ε, εφευρέθηκε το καλοκαίρι σε σχέση με ε, όσα ήταν ήδη γνωστά. Αν δείτε τα κείμενα, όλα τα κείμενα που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα διαπιστώσετε ότι είναι πλήρης η ταύτιση και ε, η εξίσωσή τους, οπότε δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Ο κύριος Βαν Ρόμπεϊ πέντε φορές προείδρευσε στο Eurogroup σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ε, γιατί ο κόσμος απορεί και εξίσταται επειδή συνεδριάζουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και ε, προεδρεύει ο κύριος Βαν Ρομπέι. Προτιμώ να είναι εκείνο παρά κάποιο άλλος. Ο Χέρμαν προεδρεύει και τους 27. Γιατί να μην μπορεί να προεδρεύσει στους 17. Δεν κατάλαβα. Αξιόπιστη οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη μπορεί να συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και ως Δεμαγίας ε, έμπλεος θαυμασμού ο υπόλοιπο κόσμος θα γονάτιζε και θα υπογλιόταν σε μια εξαμηνιαία συνεδρίαση. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σε επίπεδο ε, προζώνης να δίνει ε, προσανατολισμούς, να δίνει κατευθυντήριες γραμμές και να λειτουργεί σωστά με τη δόση αντίδραση που χρειάζεται. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι ο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών δεν θα γίνεται μετά το Eurogroup σε επίπεδο κρατών και κυβερνήσεων. Αντίστροφα, πρώτα στις εθνικές πρωτεύουσε και να λένε όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών τα ίδια με τους Πρωθυπουργού και όταν ομιλεί ο Πρωθυπουργό ο εκάστοτε να εκφράζει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία στην οικονομική διακυβέρνηση, οικονομική κυβέρνηση, διάβασα καμιά εκατοστή διαφορετικέ εκδοχές αυτή τη βδομάδα και μισές ήταν στα γερμανικά. Σα ευχαριστούμε. Στρέφομαι ευθύ αμέσω προς τον Επίτροπο Ρένε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σε 5-6 λεπτά θα αποχωρήσουν οι διερμηνείς. Βιαστείτε παρακαλώ. Ευχαριστώ, Σάρων. Σας ευχαριστώ όλους ε, γιατί ήταν, η συζήτηση χαρακτηρίζεται από μεγάλη υπευθυνότητα και αυτό απηχεί και την σοβαρότητα της προϊούσας ε, κρίσης ε, που πλήττει την ευρωπαϊκή οικονομία και την απασχόληση. δεν μπορώ να δώσω επιμέρους απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μπορώ να σχολιάσω κάποια από τα πιο σημαντικά ζητήματα. για τις χώρες για τις οποίες ζητήσατε περισσότερες πληροφορίες και κάνατε ερωτήσεις. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ε, κάνουμε την αναθεώρηση των ε, εθνικών προγραμμάτων για την Ελλάδα, για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία μεταξύ άλλων και εν ευθέτω χρόνο θα επανέλθω στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ε, σύντομα για να κάνουμε ενδελεχή συζήτηση για αυτά αν κρίνεται ότι είναι σκόπιμο για τις δικές σας εργασίες. Πιστεύω ότι αυτή είναι η βάση για να αποκαταστήσουμε την οικονομική βιωσιμότητα και να έχουμε τις ε, απαιτούμενες προϋποθέσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να ακολουθηθούν αυτά τα προγράμματα και να βοηθούν τα εθνικά προγράμματα της χώρας ε, να σημειώνουν πρόοδο. Ε, χρειαζόμαστε ένα μακροπρόθεσμο όραμα, είπαν κάποιοι και θα συμφωνήσω. Είναι σίγουρο αυτό και στην τωρινή συγκυρία θα πρέπει να εργαστούμε σε πολλά μέτωπα και με όλες τις ε, ε, χρονικές προοπτικές ε, αν θέλετε γιατί τα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα θέματα είναι αλληλένδετα θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για την αντιμετώπιση της τωρινής κρίσης και παραλλήλου να εργαστούμε ούτως ώστε η αρχιτεκτονική της οικονομικής πολιτικής μας να γίνει πιο εύρωστη, πιο κρατεά. Και από αυτή την πλευρά έχει τόσο μεγάλη σημασία η δέσμη των έξι οδηγιών και απευθύνω έκκληση και προς το Συμβούλιο και προς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιολογήσουμε τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, ναι μεν, αλλά ταυτόχρονα αυτή η δέσμη έχει και βραχυπρόθεσμη επιρροή ως προς την εμπιστοσύνη των αγορών και καταδεικνύει τη συλλογική μας ε, ικανότητα να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κρίση και να δημιουργήσουμε ερίσματα για περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία και τόνωση της απασχόλησης. Επίση, έχει συγκεκριμένη επίδραση ω προ των ε, πολιτικών που θα ακολουθήσουμε σχετικά με την δημοσιονομική βιωσιμότητα αλλά και τα νέα μέσα ε, του οικονομικού ε, συντονισμού. Θα ενθαρρύνουμε επίσης τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πολιτικές για να τονώσουν την ανάπτυξη και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και είναι η ουσία τη ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Ε, θα συμφωνήσω με αυτούς που είπαν ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα, να έχουμε το μακροπρόθεσμο όρεμα, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε για να υπερπηδήσουμε τις βραχυπρόθεσμες ε, προκλήσεις. Και από αυτού θα έλεγα ότι καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε ένα κατά τα άλλα γνωστό πρόβλημα. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εργάζονται σε μικροδευτερόλεπτα με αυτή την ταχύτητα, ενώ η δημοκρατία, η πολιτική ε, κινείται ε, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε δεκαετία. Ε, και όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό, για να μεριμνήσουμε ώστε ε, μια δημοκρατική πολιτική να ε, δείξει το δρόμο στις αγορές. Πρέπει ε, να φροντίσουμε ώστε οι δομές που έχουμε να είναι ευφιέστερες, θεμητότερες και να πλαισιώνουμε την λειτουργία των αγορών. Επίσης θα πρέπει να δούμε και με το να επανεξετάσουμε μάλλον τον τρόπο λειτουργία των θεσμικών μα οργάνων και συγκεκριμένα τη Ευρωζώνης και των διαφόρων συνθέσεων που υπάρχουν ε, στην ζώνη αυτή. Έχουμε κοινή ευθύνη για την ζώνη ευρώ και ε, ε, ξεχωριστή επιμέρους ευθύνη για κάθε ένα κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να τονίσω επίσης ε, τη βραχυπρόθεσμη ανάγκη για να ληφθούν ε, αποφάσεις που θα έχουν όμως και μεσοπρόθεσμη ε, επιρροή. Όχι μόνο οι δέσμοι των έξι οδηγιών, ούτε και μόνο η απόφαση που ελήφθη την 21η Ιουλίου στη Σύνοδο για τις χώρες της Ευρωζώνης. Όλες οι αποφάσεις που θα ληφθούν αποτελούν την βάση της μελλοντική λύσης για την κρίση και ε, επ' αυτού θέσατε στις διάφορες ερωτήσεις για να ενισχύσουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη προς την ευρωπαϊκή οικονομία. Εργαζόμαστε τώρα άοκνα ώστε η συμφωνία της 21ης Ιουλίου να υλοποιηθεί τάχιστα. Ε, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένες της συγκυρία της αυξανόμενης αβεβαιότητας και ε, διαρκούς επιβράδυνσης της οικονομικής πορείας σε παγκόσμιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ας πω και κάτι θετικό. Ε, διάφορα κράτη της Ευρωζώνης ε, έχουν επισπεύσει τις εθνικές διαδικασίες ε, επικύρωσης και βελπιστώ, είμαι μάλλον πεπισμένος ότι μέχρι τα τέλη, μέσα ή τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει περατωθεί η διαδικασία, υπερατωθει η διαδικασια αυτα σε πρόθεσμο επίπεδο, δηλαδή με επικύρωση και εφαρμογή της Συμφωνίας 21η Ιουλίου. Ας το κάνουμε αυτό και μετά περνάμε στην επόμενη φάση της οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης. Ρωσίας. Εν κατακλείδη θα έλεγα ότι ε, όσο πιο γρήγορα θα διευκρινίσουμε τα επιμέρους στοιχεία αυτής της συμφωνίας, τόσο περισσότερο θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη όλων ε, προς εμάς, ε, δηλαδή προς την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε την κρίση σχετικά με την διαφωνία για τις εγγύησεις. Λοιπόν, θα πρέπει να διεκπαιρεωθεί ταχύτατα και η Επιτροπή θεωρεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να έχει κρατεά νομική βάση πρώτον. Δεύτερον, να χαρακτηρίζεται από συνέπεια σε σχέση με ε, τα ε, ε, χρηματοπιστατικά προγράμματα, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και τα επιμέρους προγραμμάτων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συγκεκριμένα στην περίπτωση της Ελλάδας. Και τρίτον, θα πρέπει η λύση να υποστηρίζεται από όλα τα μέλη της Ευρωζώνης, από πλευράς μας, από πλευρά δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διευκολύνουμε τη διευθέτηση αυτού του θέματος στις, σε διαπραγματεύσεις με όλα τα μέλη της Ευρωζώνης ε, με τρόπο ώστε ε, να επιτύχουμε ε, ταχεία και ορθή εφαρμογή της συμφωνίας της 21 η Ιουλίου. Οι, μέσο, οι μεσοβραχυπρόθεσμες προκλήσεις αυτές είναι. Ας περιμένουμε λοιπόν να περατωθεί η διαδικασία και μετά θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για την οικονομική διακυβέρνηση και για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι έχουμε και άλλη συνεδρία προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Ευχαριστώ.